Okay, colleagues. There's another thing. καθώς ξεκινάει η συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφη, θα ήθελα να καλωσορίσω τον εμπορικό επιμελητήριο της Δυτικής Πομερανίας, εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο που έχει προσκαλέσει ο κύριος Κούνε. Καλώς ήρθατε εδώ και ελπίζω να σας ε, τραβήξει ενδιαφέρον η συνεδρίασή μας. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Is everybody happy with the agenda? Η ημερήσια διάταξη πρακτικά 18-19 Μαρτίου, 25-26 Μαρτίου εγκρίνονται καλώς. Στη συνέχεια έχουμε την αναφορά. Έχουμε την γνωμοδότηση τη δική μου. για τους κανόνες φοιτικούς με τις κρατικές ενισχύσεις προτείνονται αλλαγές στο σχετικό κανονισμό για τις μεταφορές σιδηροδρομικές και οδικές και με ανησυχεί ιδιαίτερα στη διαδικασία που έχει επιλέξει για την τροποποίηση του κανονισμού 1370 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το λεγόμενο κανονισμό πρόσδοσης εξουσίας για τις κρατικές ενισχύσεις. Το άρθρο 9 της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής του εν λόγω κανονισμού ε, πάβει να ισχύει έξι μήνες μετά την θέση σε λειτουργία του κανονισμού που υιοθετείται ε, σε σχέση με την κατηγορία αυτή των κρατικών ενισχύσεων. Το εν λόγω άρθρο αποκλείει από την υποχρέωση της, πρώιμης, της πρώτερης ε, κοινοποίησης τις υπηρεσίες TFU σε σχέση με τη μεταφορά των επιβατών με βάση της ε, ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τον κανονισμό αυτών. Η αλλαγή αυτή λοιπόν σε σχέση με τον κανονισμό 1370 που μπορεί να προκύψει με τον κανονισμό πρόσδοσης εξουσίας καθιστά πολύ δυσβάσταχτη και ε, ενοχλητική αυτή την πρόταση. Ο κανονισμός είναι νομοθετικό κείμενο, υιοθετήθηκε από την κοινή νομοθετική διαδικασία και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτο για μένα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση ενός κειμένου που προκύπτει από ε, την νομοθετική διαδικασία με μόνη από ένα μη νομοθετικό συμβούλιο, από ένα μη νομοθετικό κανονισμό ε, με μόνη τη διαβούλευση του Κοινοβουλίου και τι θα έπρεπε να απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει σχετικές προτάσεις κατά τρόπο της κοινής νομοθεσίας. Επιπλέον, μια νέα πρόταση που υιοθετείται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συμπεριέλαβε τις εν λόγω προτάσεις του κανονισμού πρόσδοση ε, αρμοδιοτήτων δηλαδή. Γιατί δεν περιλήφθησαν στην πρώτη αυτή τακτική νομοθετική, τακτικής νομοθετικής διαδικασίας τροποποίηση. Έτσι λοιπόν με το σχεδιασμό της προτάσεως για, την, ε, για τον κανονισμό πρόσδοσης εξουσιών ε, αρμοδιότητας προφανώς παραβλέπει τις νομοθετικές εξουσίες και προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό θα έπρεπε εφόσον το επιθυμούσε η Επιτροπή, να έχει περάσει μόνο από την τακτή νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή των Οικονομικών Θεμάτων έχει τη ουσία αρμοδιότητα. Εμείς ε, δυνάμει το άρθρο 5 όσον αφορά τις δικές μας ε, αρμοδιότητες για τον ε, κάρονισμο πρόσθεση που αφορά τις δημόσιες ε, μεταφορές μόνο έχουμε γνωμοδότηση, αλλά δεδομένων των εξέλιξεων στο Συμβούλιο, γιατί έχουν δεχθεί, μια πρόταση από την Ιρλανδική Προεδρία τα κράτη, όπου διαγράφεται κάθε αναφορά στον καρονισμό PSO και με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει και τις διαβεβαιώσεις τόσο της Προέδρου και του εισηγητού, ότι δηλαδή θα προσπαθήσουμε να, κάνουν, να εξασφαλίσουν απάλληψη των σχετικών διατάξεων του κανονισμού PSO, πιστεύω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την διαδικασία του άρθρου 49 για τη γνωμοδότηση. Υπενθυμίζω στην Επιτροπή μα ότι για να παρακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή των Οικονομικών πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα στην έκδοση αυτή τη νομοδότηση. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι πολύ στενό τα χρονικά περιθώρια. 25 Απριλίου το μεσημέρι στις 12 θα έχουμε την προθέση για την κατάσταση των τροπολογιών, οι οποίες μπορούν να κατευθούν μόνο στα αγγλικά, ιδάλλως δεν θα προλάβουμε τους ρυθμούς της Επιτροπής των Οικονομικών. Το σχέδιο γνωμοδοτήσεως, το οποίο έχετε στον φάκελό σας, βρίσκεται μόνο στα αγγλικά, δεν έχει μεταφραστεί ακόμη, αλλά φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε πως η γνωμοδότησή μου θα περιοριστεί σε μία μονοτροπολογία, με μία μόνο λέξη, διαγραφή της εν λόγω προτάσεως από το άρθρο 9. Δεν θα είναι λοιπόν μακροσκελής η γνωμοδότηση. Μόνο μία τροπολογία, η οποία θα λέει μόνο delete για το άρθρο 9, διαγραφή. Μία λέξη. Καταλαβαίνω βέβαια ότι δεν είναι αυτό όπως ε, θα θέλαμε, το να πρέπει δηλαδή να δουλεύουμε, πάντα, ε, να δουλεύουμε μόνο στα αγγλικά με το κείμενο αυτό, αλλά εφόσον πρέπει να προλάβουμε την Επιτροπή των Οικονομικών, Επαναλαμβάνω λοιπόν προθεσμία για κατάθεση τοπολογιών 25 Απριλίου και ελπίζω ότι θα έχετε στα αγγλικά την έκθεσή μου και θα δεχτείτε τις θέσεις μου. Κύριος Γκρός έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ω προς το περιεχόμενο καταρχάς. Συμφωνούμε απολύτω και εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο δεν πρόκειται να καταθέσω τροπολογία. Πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 2, λέει ο μιλητή. Όπω και ο εισηγητή, διερωτώ με και εγώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια πρόταση με βάση τον κανονισμό πρόσδοση εξουσία, ενώ είχε ήδη μέσα από τη διαδικασία της, ε, την τακτική νομοθεσία, την νομοθετική, ε, διαδικασία την νομοθετική, τη δυνατότητα να εισαγάγει τι σχετικέ τροποποιήσει. Δεν ξέρω καν, ε, χωρί να είμαι βέβαια νομικό, αν είναι και θεμητό ή νομητό νομικά σωστό να κάνει αυτές τις αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει όμως θα ήθελα μια εξήγηση. Γιατί η τροποποίηση του 1370 του 2007 γίνεται με αυτόν τον τρόπο που μας εξήγησε ο Πρόεδρος. Και μια τελευταία ανακοίνωση εάν τυχόν, αν και δεν φαίνεται τέτοια ε, πιθανότητα ευτυχώ. Εάν τυχόν όμω παρελπίδα συμφωνεί στο Συμβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα υπόσχομαι ότι στη δική μου την έκθεση Public Service Obligations, υποχρέωση δηλαδή για παροχή ε, δημόσια υπηρεσία, θα επανέλθει το θέμα αυτό και δεν πρόκειται να το αφήσουμε. Καλώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κύριο Σαλκαντραού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομο. Εγώ και για ομάδα προσωπώ μπορούμε να σα στηρίξουμε σε αυτό που προτείνετε, όχι μόνο για λόγου ε, τύπου, αλλά και για λόγους ουσία. Οπότε έχετε και τη δική μα υποστήριξη. Κύριο Στεμπάκα. Πολύ σύντομο θα είμαι. Για μένα η αναρμόνιση, ο εξυγχρονισμός είναι μια καλή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά έχω και εγώ τις ίδιες παρατηρήσεις και τις ίδιες ερωτήσεις που ακούσαμε όσον αφορά την νομοθεσία. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που κάνατε εσείς πάντως για το πακέτο αυτό. Είναι καλό αν τελικά πάει κάτι στραβά να μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Και έχω και μια ερώτηση προς εσάς όσον αφορά το άρθρο 1 εξ, ε. Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι οι λόγοι. Κατά τα άλλα πάντως είμαι και εγώ στην ίδια γραμμή με εσάς. Κύριος Ναι, και δική μου ομάδα υποστηρίζει την θέση σας πλήρως έχουμε την ίδια, τις ίδιες ανησυχίες με σένα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υποτροπιάζει. Και διαρωτώ με τι έχει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ύστερα από δύο χρόνια με τα Giga Liners βλέπει ότι δεν μπορεί να κάμψει τη θέλησή μας και ενώ είναι θεματοφύλακας των συνθήκων και της νομοθεσίας προσπαθεί να τις ανατρέψει, να ανατρέψει την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται και ενώ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία τακτική ε, νομοθετική διαδικασία έρχεται με την παράνομη μέθοδο να εισαγάγει μια ε, τροποποίηση. Εδώ μιλάμε για ανατροπή μιας νομοθετικής διαδικασίας, την οποία το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο από κοινού έχουν επεξεργαστεί και εγκρίνει. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν, σε ποια παράγραφο, ποια συνθήκη και ποιο άρθρο ε, αναφέρεστε για να προχωρήσετε με αυτή τη μέθοδο. Πολύ καλά ε, λέει ο κύριο ε, Γκρό ότι αν ε, τυχόν δεν τα καταφέρουμε θα βρούμε και άλλη λύση. Αλλά όχι, δεν πρόκειται να χρειαστεί άλλη λύση. Η ίδια διαδικασία όπω και την άλλη φορά θα καταθέσουμε μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά ένα θεσμικό όργανο προσπαθεί να παραγκονίσει το Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε κάθε δυνατή πρωτοβουλία. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, αλλά πιστεύω ότι και εσύ ω πρόεδρο τη Επιτροπή για άλλη μια φορά θα πρέπει να καταγράψει και να δηλώσει την δυσφορία μας ως προς τις διαδικασίες αυτές οι οποίες είναι απαράδεκτες και εν πάση περιπτώσει αύριο που θα είναι εδώ ο Επίτροπος καλό θα ήταν να εξηγήσει τι είδους νοοτροπία και λογική είναι αυτή η οποία τον οδήγησε στο να παραβιάζει το δίκαιο αντί να το προστατεύει. Ευχαριστώ που κύριε Κράμερ. Πρέπει να πω ότι με καταλάβανε ή τουλάχιστον έχω εκφράσει αρκετά ξεκάθαρα τις θέσεις μου. Ο κύριος Ζέλαρ. Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να κρύψω ότι θα υποστήριξω και εγώ τις δικές σας θέσεις. Δεν είναι οι διαδικασίες αυτές ε, νόμιμες ή φυσιολογικές. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει μάλιστα γιατί και τι ε, διεκδικεί, τι προσπαθεί να, τι επιδιώκει με αυτή τη ε, διαδικασία που έχει επιλέξει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρίκε δεν θέλει το λόγο. Από την Επιτροπή. Κυρία Μερσέντες Κάμπο, έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να σε εξηγήσω καθαρά τα νομικά επιχειρήματα που ήταν η βάση της πρότασης της Κομισιόν. Καθαρά νομικά επιχειρήματα, παραλαμβάνω. Ο Κασνός 1370-2000 ε, ε, είναι ο κανονισμός για τις μεταφορές και προσαρμόστηκε ε, στα δεδομένα μια διπλή νομική βάση το κείμενο άρθρο 91 τη συνθήκη που είναι η νομική βάση για τι μεταφορέ και το άρθρο 190 της συνθήκης που επιτρέπει στο Συμβούλιο να ορίσει τους συγκεκριμένους κανόνες συμβατότητας για τις ενισχύσεις εκείνες που δεν χρειάζεται να κοινομηθούν στην Κομισιόν. Για αυτό το κανονισμό και τις μεταφορές, εδώ έχουμε την περίπτωση του άρθρου 9 που πρώτα απ' όλα μιλάει για τις δαθμίσεις στις υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας εισήχθη ένα νέο άρθρο, το άρθρο 108 παράγραφος 4, το οποίο εισάγει μια νέα πρόχρηση, αν θέλετε, σε αυτό το κανόνα και δίνει στην Κομισιόν πλέον την αποκλειστική αρμοδιότητα να ορίσει τους συγκεκριμένους αυτούς κανόνες συμβατότητας για αυτές τις κατηγορίες ενισχύσεων που δεν απαιτείται να κοινοποιούν τις Κομισιόν. Η Κομισιόν δηλαδή σε συμφωνία και με το Κοινοβούλιο με βάση το άρθρο 109 το οποίο παραμένει απαραλλακτό μπορεί να ορίσει τις γενικές αυτές κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να εξαιρεθούν από την κοινοποίηση Μόνο η Κομισιόν είναι αυτή που ορίζει τις λεπτομέρειες, δηλαδή τους όρους συμβατότητας. Ο κανονισμός 1370 είναι υπό επανεξέταση αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια βράση Κομισιόν για την εισαγωγή κάποιων τροποποιήσεων στους κανόνες του κανονισμού. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε παράλληλα το κείμενο άρθρο 9 διότι έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και μια νέα δέσμη κανόνων ενισχύει. Γι' αυτό το λόγο και μόνο η Κομισιόν πρέπει να προτείνει την εισαγωγή του άρθρου 9 στον εφαρμοστικό κανονισμό ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν μπορεί να παραμείνει η δυνατότητα το Συμβούλιο να είναι εκείνο που θα ορίζει τι λεπτομέρειε. Η Κομισιόν πλέον έχει αυτή την αρμοδιότητα βάσει τη συνθήκη Λισαβόνα. Γι' αυτό πρέπει αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα εξαίρεσης ε, από κοινοποίηση για αυτές τις ενισχύσεις δημόσιων υπηρεσιών, να κάνουμε αυτή την αλλαγή στον κανονισμό. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αλλάξει η ουσία του άρθρου 9 είναι καθαρά μια νομική διευθέτηση, νομική αναγκαιότητα, αν θέλετε, ώστε το παράγωγο δίκαιο να ευθυγραμμιστεί με το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ξεκαθάρισα κάπως τα πράγματα. Well, I... Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Τώρα δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος αν το κάνατε αυτό, αλλά σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση όταν ακούω όρους όπως νομική αναγκαιότητα, αρχίζω και υποψιάζομαι τα πράγματα εγώ ως αιρετός, εδώ εκπρόσωπος των Ευρωπαίων πολίτων. Ε, έτσι βλέπω σαν είναι ένα τέχνασμα να μείνει εκτός εθικασίας στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπράτμαν παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περίμενα να πάρω το λόγο. Ήθελα να ακούσω την Επιτροπή, τον Επίτροπο βασικά. Τώρα ακούμε για τον άρθρο και για το άλλο άρθρο. Καταλήγει στο θέμα της διαφάνειας όμως. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν εμείς ως Κοινοβούλιο δεν εμπλεκούμε στο ίδιο το θέμα, το οποίο όπως υπενθύμησαν και άλλοι από προηγούμενες συζητήσεις, τους αρχικούς κανονισμούς που κάναμε για τις κρατικές ενισχύσεις κλπ, είναι μέτρα ιδιαίτερα επίμαχα. Γι' αυτό το θέμα δεν είναι μόνο η νομική θέση, είναι το θέμα της λογικής θέσης. Τι δηλαδή τελικά είναι πιο λογικό και πρέπει να συζητήσουμε εμείς που είμαστε το εκλεγμένο σώμα των ευρωπαϊκών οργάνων είτε πρόκειται για συμμόρφωση με το ένα με το άλλο άρθρο, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαστε ανοιχτοί και να μπορούμε να συζητήσουμε την πρόταση, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως Πρόεδρε, αυτό είναι το σωστό και πρέπει να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε εμείς που είμαστε εκλεγμένοι πολιτικοί να συμμετέχουμε, γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για νομικίστικα θέματα, είναι και θέμα ουσίας. Ευχαριστώ κύριε Λεγεπέρια. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Δύο λόγια Εάν υπάρχουν αναγκαιότητε, νομικέ αναγκαιότητε, legal necessities, θα πρέπει και να τηρηθεί το legal necessity τη κοινοβουλευτική διαδικασία. Μην φτάσουμε δηλαδή με το αλάφτον του Πάπα να αποφασίζουμε και να εισάγουμε νέες ερμηνείες. τα νομοθετικά κείμενα ε, χαρακτηρίζονται από το γεγονό ότι τα προηγείται αυτό μια, νομοθετική, μια νομοθετική κοινοβουλευτική διαδικασία. Το legal necessity σημαίνει απλώ. Ε, να προσπαθεί κανείς να είναι καθολικότερος του Πάπα. Και μια και δεν είμαστε στην Καθολική Εκκλησία. Αλλά σε ένα κοινοβούλιο, καλό τους πάντες να ακολουθήσουν τον συνήθι νομοθετικό ε, δρόμο. Αυτό το λέω και ως μέλος της Επιτροπής των Νομικών Υποθέσεων. Κύριος Κράμερ. Η νομική μας υπηρεσία ήδη έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θέλετε να ρωτήσουμε, να τα πούμε πάλι στην Επιτροπή, να ρωτήσουμε το γερμανικό Bundestag που έχει και πιο πολύ εμπειρία. Ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι μαγειρεύεται στο Bundestag. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι οι νομικές μας υπηρεσίες συμμερίζονται τις απόψεις μας. Δηλαδή έχουν ερμηνεία διαφορετική από αυτήν της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής. Φαίνεται να υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις απόψεων μεταξύ νομικών υπηρεσιών αυτή την εποχή. Λεγεμένα, όπω πολύ σωστά επισημάνει ο κ. Μπράτσμορ, το ζήτημα είναι ότι η υπηρεσία τη δημόσια υπηρεσία, τη δημόσια μεταφορέ, συνιστά και κέριο στοιχείο τη δημόσια υπηρεσία και κυρίω για τα αστικά κέντρα και τι πόλεις μα. Και ω εκ τούτου το να βγει ο κανονισμό που διέπει αυτό το ζήτημα τον, ο 1370 δηλαδή και να υπαχθεί σε μία πράξη εξουσιοδότησης χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίε που προβλέπουν την ε, συμμετοχή στο κοινοβούλιο, του Κοινοβουλίου σε αυτήν την νομοθετική διαδικασία και χωρί καν να προσδιορίζεται, να έχει προσδιοριστεί προηγουμένω τη συνιστά αυτή τη δημόσια υπηρεσία, είναι επικίνδυνο και αντισυνταγματικό ε, όποια συνθήκη και να επικαλεστεί κανεί. Λόγω του ρόλου που έχει να διδραματίσει το Κοινοβούλιο σε αυτέ τι υποθέσει. Και για να είμαστε πολύ ειλικρινεί, η παροχή δημόσια υπηρεσία από τι δημόσιε μεταφορέ ε, στο ζήτημα, το να υπάγεται στις κρατικές ενισχύσεις, πραγματικά μου γεννά μεγάλη δυσφορία και ενισχύει. Ακριβώς γιατί πρόκειται για δημόσια υπηρεσία. Άρα λοιπόν προτείνω να διαγραφεί ή κολλάβει και νομικοί μπορούν να το συζητάνε όσο θέλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι αυτή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος για το πιεσό. Δεύτερον, παραγκονίζει το κοινοβούλιο και ως εκ τούτου και για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Γκρός Μια παρατήρηση, όχι, όχι ερώτηση, πρόταση ίσως. Μήπως κύριε Πρόεδρε θα ήταν δυνατόν και να εκφράσετε την επιθυμία μας ότι το ζήτημα αυτό της ε, κινητικότητας θα έπρεπε να παραμείνει στη Γενική Διεύθυνση για τις μεταφορές τη MOVE. Έτσι ώστε να έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν και την υπόθεση και τη σημασία πάνω από όλα αυτών των πτυχών. Αλλά και διότι δεν πρόκειται για τρέχοντα ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Δεν είναι απλά δηλαδή τα πράγματα όταν πρόκειται για δημόσιες μεταφορές. Που λέτε στην περίπτωση αυτή. Μιλάμε για ένα θύμα ουσιαστικά ανάμεσα σε αυτόν τον ιστορικό πόλεμο, ανάμεσα στην Κομισιόν και κατανοώ αυτό που λέτε. Εγώ δεν, δεν με νοιάζει. Ας έχουν αφεντακτική, αλλά όταν τελικά βγουν από αυτό τον κύκλο οποίο έχουν, στον κυκαιώνα στον οποίο έχουν μπλακεί, τελικά να δοθούν αυτά που αναλογούν στο κοινοβούλιο. 25 Απριλίου καταληκτική ημερομηνία τη τροπολογία. Συμφωνείτε με τη δικασία. Ξέρω ότι είναι μόνο στα αγγλικά, θα είναι ταχύτερη διαδικασία, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι συμφωνείτε όλοι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας σε αυτό το θέμα και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης και αφορά την αφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία η συγγήτρια η κυρία Ντε Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 απέκτησε μια αποτελεσματική νομοθεσία όσον αφορά την έρευνα αεροπορικών ατυχημάτων. Σήμερα όμως φαίνεται ότι πρέπει να υιοθετήσουμε νέους κανόνες για να ενισχύσουμε την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων. Στόχος λοιπόν τη πρόταση αυτή είναι ακριβώς να πάρουμε μαθήματα από τα ατυχήματα που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά ατυχήματα, να τα προλάβουμε. Δυστυχώς ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη καταστροφή. Κάτι το οποίο το έχουμε δει στις αεροπορικές καταστροφές, ότι είναι συνδυασμό αιτιών. Γι' αυτό και το 2003 βάλαμε τις βάσεις για μια νομοθεσία η οποία θα επέτρεπε στους πιλότους ή και στους ελεκτές ενέωρια και κυκλοφορίας να αναφέρουν από μόνοι τους ένα συμβάν κάτι, ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τέτοια δεδομένα και να αποφύγουμε μελλοντικά ατυχήματα. Μετά από αρκετά χρόνια ε, φάνηκε ότι κάπως περιορίζεται το εύρος των αποτελεσμάτων αυτής της οδηγίας και γι' αυτό και θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σήμερα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να αποφεύγουμε ατυχήματα είναι να συλλέγουμε πληροφορίες όσον αφορά ε, συμβάντα που έχουμε στον ανέριο χώρο. Και για να συλλέγονται τα δεδομένα αυτά πρέπει το προσωπικό το οποίο εντοπίζει την ύπαρξη ενός συμβάντος, κάποιο λάθος για παράδειγμα το οποίο έχει κάνει ο ίδιος, να μπορεί να το κοινοποιεί από μόνος του. Άρα λοιπόν ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί και τη βάση του συστήματος αυτού. Και αυτό σημαίνει, εκτός βέβαια αν έχουν προβεί σε κάποιο πολύ σοβαρό ε, παράπτωμα, ε, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται από την ιεραρχία επειδή αναφέρουν το συμβάν αυτό. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή εμπιστοσύνη, αυτό που λέμε η κουλτούρα του δίκαιου. Πάρα πολλά συμβάντα αναφέρονται σε διάφορες χώρες από οργανώσεις ή υπαλλήλου. Ε, οι υπάλληλοι αυτοί λοιπόν όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν τέτοια συμβάντα χωρίς να φοβούνται τιμωρία. Ο μόνος στόχος αναφοράς αυτής είναι να συνεισφέρουν στην αποφυγή νέου τέτοιου συμβάντος και ενδεχομένως ατυχήματος. Η διάρθρωση τώρα, ασφάλεια, ενέργειας και δικαιοσύνη είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συνδέονται χωρίς προβλήματα και αυτό είναι και το βασικό στην πρότασή μας. Οι δράσεις αυτές πρέπει να βασίσονται στην ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη. Αν ένας υπάλληλο απολυθεί επειδή κοινοποίησε ένα τέτοιο συμβάν, κάτι το οποίο βέβαια αντιβαίνει στην νομοθετική αυτή πρόταση, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα μηχανισμό ε, προσφυγής, να μπορεί να προσφύγει δηλαδή και να καλυφθεί από το μηχανισμό αυτό, δεδομένου ότι απλώς ανέφερε αυτό το συμβάν. Έπειτα πρέπει να δούμε και το θέμα της σοβαρής αμέλειας, έτσι ώστε να μπορούν να τυχαίνουν τις ίδιας κάλυψης όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι αναφέρουν κάποιο συμβάν. Αναφέρονται διάφορες σκέψεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο πέρα, προκειμένου να έχουμε έτοιμο αυτό το περιβάλλον εμπιστοσύνη μέσα στο οποίο θα κινούνται οι υπάλληλοι. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο το οποίο προτείνεται εδώ είναι επαρκές. Έπειτα, συλλογή πληροφοριών σίγουρα αποτελεί τη βάση. Μετά πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε για να προλάβουμε νέα ατυχήματα. Εδώ συμφωνούν όλοι για το ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγουμε και να υπάρχει ένα προδραστικό σύστημα αποτελεσματικό, άρα οι διάφορες αρχές πρέπει να αναλύουν τα δεδομένα και να εντοπίζουν ε, σημαντικά σημεία. Έπειτα η ασφάλεια έχει κάποιο τίμημα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια. Αν αποφασίσουμε να ξαναδούμε τους σημερινούς κανόνες για να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, τότε εμείς οι ευρωβουλευτές πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Δηλαδή να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται, αλλά μετά να γίνεται και αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων αυτών. Για αλλιώ όλες αυτές οι προσπάθειες πάνε στράφη. Έπειτα η προβληματική της ασφάλειας ε, δεν περιορίζεται βέβαια στα σύνορα μιας χώρας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, οπότε η ανάλυση αυτή των δεδομένων πρέπει να γίνεται πάρα πολύ καλά, άρα να ενισχυθεί η ανάλυση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΣΑ η οποία έχει ένα κεντρικό ρόλο εδώ, πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Έπειτα η νομοθεσία. Η νομοθεσία λέει ποια είναι τα συμβάντα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται. Και έχουν την υποχρέωση δηλαδή οι υπάλληλοι να αναφέρουν. Και εδώ θέλουμε να προσθέσουμε και αυτά τα οποία κρίνουν σε θελοντική βάση ότι θα ήταν καλό να αναφέρουν. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια νομική πλαισίωση. Είναι δύσκολο να δώσουμε έναν κατάλογο παραδειγμάτων, αλλά θα έπρεπε παρόλα αυτά να δώσουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο για να ξέρει ο καθένα τι δηλώνει, τι αναφέρει. Το πεδίο εφαρμογή να είναι συγκεκριμένο, όπως λέω και στην ε, έκθεσή μου, ακόμα και για τα σκάφη αναψυχή, τα πιο μικρά αεροσκάφη. Ίσως δεν ε, πρέπει να έχουμε τον ίδιο κατάλογο για αυτά τα μικρά αεροσκάφη όπως και για τα μεγάλα. Πάντως ο κατάλογος θα πρέπει να είναι πλήρης αλλά προσαρμοσμένος. Όλοι ξέρουμε ότι σε ένα πλήρη κατάλογο πάντα μπορεί να ξεχάσουμε κάτι. Οπότε αν στη εθελοντική βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και αυτά τα ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι αρμόδιες αρχές, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ γιατί έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο πλήρη στοιχεία και να μπορούν όλοι να ενημερώνονται. Χρειάζεται ένα δυναμισμό το σύστημα αυτό. Να μπορούν για παράδειγμα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι, οργανώσεις ή όσοι αναφέρουν κάποιο συμβάν κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έπειτα, η πρόταση κανονισμού πρέπει να επιτρέπει και στα κράτη-μέλη και στην ΕΑΣΑ να ανταλλάσσουν τα δεδομένα. Για να πάρουμε ένα παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν μια χώρα μέλος να μην ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια για ένα συμβάν το οποίο έχει λάβει χώρα στο δικό του ενέριο χώρο, επειδή το αεροπλάνο προέρχεται από άλλη χώρα μέλος. Το βασικό πάντως είναι να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και πλήρη προς όφελος της ασφάλειας των επιβατών. Ελπίζω η σημερινή ανταλλαγή απόψεων να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε περισσότερο και να δούμε τι πράγματα πρέπει ενδεχομένω να προσθέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Λαγκτράβη, παρακαλώ, έχει το λόγο. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κ. ο ε, δεν μπορούσε να παρόν σήμερα, οπότε θέλω να πω κάποια λόγια και εξ του και εξ ονόματος της ομάδας Θέλουμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την ε, εισηγήτρια, την κυρία Τεγράκα, για την πολύ καλή τη δουλειά. Πολλά είδη η οποία ε, επισημάνονται στην χρηματοδότησή τη και ιδίω ε, η δημιουργία μια ε, καλή κούλτουρα, αν θέλετε, στον τομέα αυτό, ώστε οι αναφορέ ε, του προσωπικού να μην συνεπάγονται και τιμωρεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα τα θέματα της ε, σοβαρής αμέλειας όπως ανέφερε η συγγήτρια. το feedback για όσους κάνουν αυτή την αναφορά επιστατικών ώστε να βλέπουν και το όφελος ε, της αναφοράς που έχουν υποβάρει είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βεβαίω υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που δεν ε, ε, τα αντιμετωπίζει επαρκώς ε, στο κείμενό της συγγήτρια. Θα αναφέρω δύο. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι η πρόταση της Κομισιόνα αγνοεί πρακτικές της ΕΑΣΑ που ήδη υπάρχουν, όπως το σύστημα αναφοράς περιστατικών όπως ορίζονται, στον κανονισμό 15 και στον ε, κανονισμό 216 και τους εφαρμοστικούς σχετικούς κανόνες έχω την αίσθηση ότι κάπως έχει αγνοηθεί σε έναν βαθμό η σε αυτό το κείμενο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε υποστήριζε τη σύσταση της ΕΑΣΑ ως κεντρική υπηρεσία για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Αεροπλοεία. Και καλό λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη είναι αυτού του κανόνε. Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη την ΕΑΣΑ σε όλα τα επόμενα μέτρα και να δοθεί ευκαιρία σε αυτή να βοηθάμε την εμπειρογνωμοσύνη της ε, τον νέο κανονισμό. Έπειτα, σε ό,τι αφορά την ε, μη εμπορική αεροπλοεία. Το πεδίο εφαρμογή καλύπτει όλα τα αεροσκάφη, χωρίς να λαμβάνει όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μη εμπορικού κλάδου, όπως ε, τις διάφορες κατηγορίες αεροσκαφών και την αεραστεχνική αεροπλοεία. Και ε, εκεί θα πρέπει να υπάρχει αναλογική προσέγγιση στην αναφορά των περιστατικών και το καθηγμό του αναλογή. Αυτό συνάδει και με την Γενικότερη στρατηγική ασφάλεια στην αεροπλοεία τη ΕΑΣΑ. Θα θέλαμε λοιπόν η να λάβει υπόψη αυτά τα σχόλια και προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία για αυτό το φάκελο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κατσίν, εκ μέρους των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε συγήτρια. Πολύ χαίρομαι που συνεργάζομαι και πάλι με την κυρία Ντεβεράκ που την γνωρίζω ως ε, η δήμονα στον τομέα υπομονετικιά και έτοιμη να ε, προχωρήσει σε ε, συμβιβασμούς. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι επικοδομητικός με την έκθεση αυτή. Αυξάνεται η νέα κυκλοφορία και γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες πρόληψης. Οι έρευνες διαφόρων ατυχημάτων πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά και να αναφέρονται όλα τα περιστατικά. Πρέπει να είμαστε προδραστικοί. Τα κράτη-μέλη, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, πρέπει να φροντίζουν για τη συλλογή των ε, στοιχείων όσον αφορά τα περιστατικά αυτά. Τώρα, εκεί που μιλάμε για την προστασία των ε, αναφερόντων, πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε σε περίοδο που δύσκολα κανείς βρίσκει δουλειά. Και από την άλλη όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να κάνουν... Οπότε, εφόσον ε, υπάρχουν ε, εταιρείε οι οποίες λένε ότι πρέπει να γίνονται οικονομίες στα καύσιμα, εμείς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ανθρώπων να τους ε, βοηθήσουμε και να αποφύγουμε να απολύουν κόσμο επειδή αναφέρει διάφορα περιστατικά. Πρέπει να είναι σαφές το τι αναφέρει κανείς, ποια είναι τα περιστατικά που αναφέρονται. Έχω μιλήσει με διάφορους και θα τους ακούσω και στο μέλλον. Σίγουρα με την εισηγήτρια θα μπορέσουμε αυτό να το αποσαφηνίσουμε πριν έχουμε τη δεύτερη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η αεροπορία πρέπει να καλύπτεται στο σύνολό της. Οτιδήποτε πετάει και μεταφέρει επιβάτες μπορεί να έχει κάποιο ατύχημα, να πέσει και να σκοτωθεί κόσμος. Δεν έχει νόημα λοιπόν να αλλάξουμε τη ρύθμιση είτε πρόκειται για μικρά αεροσκάφη ή για αερόστατα ή δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία εξαρτώνται και από την ε, δυναμική, από τον αέρα της στιγμής. Πάντως είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και με τους άλλους κοιόδες εισηγητές. Ευχαριστούμε η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντεβιράκ που είναι η εισηγήτρια. Θα θυμάται κι εσείς ότι ήμουνα εισηγήτρια εγώ στην αρχική οδηγία το 2003 και νομίζω ότι το κοινοβούλιο μας έκανε τότε πολύ καλή δουλειά. Ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που προχωρήσαμε σε υποχρεωτική αναφορά περιστατικών. μετά από την εθελοντική βάση στην οποία πολλές χώρες το κάνανε αυτό. Τώρα έχουν περάσει άλλα δέκα χρόνια και είναι σαφές ότι κάποιες χώρες μέλη δεν καταλαβαίνουν καλά τι τελικά πρέπει να αναφέρουν και τι όχι. Ενώ εγώ πιστεύω ότι είναι σαφέ και άλλοι πιστεύουν ότι είναι σαφέ, αλλά όχι όλοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, τα περιστατικά τα οποία αναφέρονται είναι δύο φορέ παραπάνω από εκείνα που αναφέρονται στη Γερμανία. Ενώ η αεροπορική βιομηχανία είναι περίπου του ίδιου μεγέθου. Έτσι και δεν θέλω εδώ να, κάνω, να επικρίνω κανέναν, ούτε Γερμανία ούτε κανέναν άλλον. Απλώ λέω ότι οι κανόνε ερμηνεύονται πολύ διαφορετικά στην κάθε χώρα. Άρα είναι πολύ καλό που η συγγήτρια το λέει αυτό και προσπαθεί να το διορθώσει. Αυτό που ακούστηκε επίσης είναι το θέμα της κουλτούρας, ότι δηλαδή πολλοί άνθρωποι φοβούνται να αναφέρουν κάποιο περιστατικό, προτιμάνε να μην μπουν τίποτα. Το καλό πάντως με την αεροπορία είναι το ότι έχουμε μέχρι τώρα καλή αναφορά περιστατικών, σε πολλές περιπτώσεις που έγιναν ατυχήματα, η διερεύνηση έγινε πάρα πάρα πολύ καλά και αυτό είναι πολύ θετικό. Τώρα όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και ο συνάδελφος Ελκαντροή που μετέφερε κάποια σχόλια, έτσι και εγώ ανησυχώ λίγο γιατί η ΙΑΤΑ βγαίνει απ' έξω. Την πρώτη φορά ε, δεν υπήρχε συμφωνήσαμε να έχουμε μια, έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας, αλλά δεν βλέπω πώς θα λειτουργήσει τελικά. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ε, διαφόρων οργανισμών Ευρώπης και αλλού. Έχουμε έτσι καλλιώς τους εφαρμοστικούς κανόνες τη ΙΑΤΑ και μετά θα έχουμε παραρτήματα. Οπότε μια αεροπορική εταιρεία δεν θα ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ή που έχουμε έναν οργανισμό ασφάλειας ή που δεν έχουμε έναν οργανισμό ασφάλειας. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το πράγμα στις διάφορες χώρες, γιατί η πολιτική αεροπορία στις διάφορες χώρες θα μπερδευτεί. Και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρόλο εδώ, αλλά κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή μπερδεύεται με διάφορα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχολείται ο οργανισμό ασφάλειας και όχι Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο, δηλαδή φοβάμαι την επικάλυψη. Έπειτα για το δίκτυο αναλυτών ασφάλειας. Αν αναφέραμε κάτι, θα έπρεπε να ήταν οι ελεγκτέ ενέργεια κυκλοφορία και οι πιλότοι. Έτσι δεν είναι. Αυτοί δεν είναι εμπειρογνώμονε, γιατί του χρειαζόμαστε του εμπειρογνώμονε να παίξουν ένα ρόλο. Ποιοι είναι τελικά. Και για την ενημέρωση και τι πληροφορίε κάπου μιλάει για τους ε, υπαλλήλους ατομικά. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει... Πρέπει, πιστεύω, μέσω, για παράδειγμα, της τήσιας έκθεσης της ΙΑΤΕ να ενημερώνεται όλος ο κόσμος. Έπειτα για το European ε, Common Risk. Και αυτό μου φαίνεται περίεργο. Η συλλογή δεδομένων Μιλάτε για μια υποχρέωση σε 30 μέρες. Ναι, αν είναι κάτι περίπλοκο μπορεί να χρειάζεται παραπάνω, οπότε είμαστε πιο ελαστικοί με την προθεσμία. Και τέλος το θέμα της θελοντικής αναφοράς περιστατικών. Είναι κάπως οξύμερο να έχουμε και υποχρεωτικό και θελοντικό. Το εθελοντικό, βέβαια ξέρουμε είναι κάτι άλλο από το υποχρεωτικό. Στο, το 1992 άρχισε να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο υπάλληλο μέσα σε μια εταιρεία πρέπει να νιώθει εμπιστοσύνη και ελεύθερος να αναφέρει κάτι το οποίο του φαίνεται ότι δεν πάει καλά. Είναι κάτι διαφορετικό από το υποχρεωτικό που θα υπάρχει ο σχετικός κατάλογος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις εταιρείες και όλες τις χώρες μέλη να συμφωνήσουν και με την εθελοντική αναφορά, γιατί είναι ένα εξαιρετικό μέτρο πρόληψης ατυχημάτων και αυτό μας ενδιαφέρει εδώ. Η εισηγήτρια υπογράμμισε όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να περιπλέξουμε υπερβολικά την ρύθμιση, να χρησιμοποιήσουμε ότι ήδη υπάρχει, οπότε θα ήθελα να το έχει υπόψη αυτό και η εισηγήτρια και η Επιτροπή παρακαλώ. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι καλό γιατί στο κάτω-κάτω όλοι το ίδιο θέλουμε να καταλήξουμε στα σωστά συμπεράσματα. Έχουμε μια πολύ καλή αεροπορία στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ιδιαίτερα υψηλέ προδιαγραφές και το προσωπικό, οι πιλότοι και οι υπόλοιποι, να νιώθουν εμπιστοσύνη και να αναφέρουν περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να προλάβουν μελλοντικά ατυχήματα. Αλλά όντως το θέμα της σοβαρής αμέλειας είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν θα μπω σε αυτό τώρα γιατί δεν ξέρω, αλλά όντως αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Λίτιμπεργκερ, συγγνώμη που δεν σας έδωσα πριν το λόγο. Ε, είναι το βρετανικό, ο Για μένα η συζήτηση είναι συναρπαστική, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ την συγγητρία η οποία έκανε την πρώτη ε, παρουσίαση του θέματος. Ε, θα ήθελα να πω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται ώστε να έχουν ένα σύστημα όσο το δυνατόν απρόσκοπτα λειτουργούν και ώστε να καταγράφονται, να προλαμβάνονται όποια περιστατικά. Πλην όμως, και αυτό το βλέπουμε και από τις έρευνες, υπάρχουν πολλοί λόγοι και διαφοροί για τους οποίους θα πρέπει και να ανησυχούμε. Ε, διαμορφώνεται ένα corpse ένα πνεύμα ομαδικό, ότι δεν θα πρέπει να καταγράφονται, να δημοσιοποιούνται περιστατικά ή το πολύ πολύ θα πρέπει να συζητούνται σε κλειστό κύκλο. Ε, εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η αλλαγή ε, νοοτροπίας, γιατί ακριβώς χάρη στη δημοσιοποίηση μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης, όταν κάποιος καταθέτει μια αναφορά και επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν θα πρέπει να βρίσκεται ή να κινδυνεύει να ρωθεί σε τη σημερινή κατάσταση, να υποστεί συνέπειε. Τώρα, εν ώψη και τη οικονομική κρίση, είναι πολύ περισσότερες οι δυνατότητες που θα είχε μια επιχείρηση να ασκήσει πίεση στον εργαζόμενό τη. πολλές φορές δεν και προληπτικά, και αυτό λογοκρίνεται ταυτόχρονα κάθε εργαζόμενος, δεν συμμετέχει, δεν συνεργάζεται στην ε, δήλωση και καταγραφή αυτών των ε, περιστατικών. Αυτό που θα πρέπει δηλαδή να προβλέψουμε θα ε, πρέπει να είναι η διασφάλιση οποιοδήποτε καταγγέλει ένα περιστατικό ε, με στόχο βέβαια πάντα την βελτίωση της ασφάλειας στις αερομεταφορές στην αέρια κυκλοφορία. δεν κινδυνεύουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι δεν θέλουμε και να αλλάξουμε τίποτα. Ε, επίσης, στην διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτικής, ε, ιδιωτικών πτήσεων κτλ. Υπάρχει ένα ψυχολογικό, ένας ψυχολογικός φραγμός γιατί ποιος ε, θα κακολογήσει ή εν πάση περιπτώσει θα καταγράψει ελάττωμα τεχνικό στο δικό του αεροπλάνο. Το βλέπουμε και με τους ε, ιδιοκτήτες φορτηγών, ότι δεν παραδέχονται ποτέ, φορτηγών ε, αυτοκινήτων εννοείται, ε, δεν παραδέχονται ποτέ ή πολύ δύσκολα κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο φορτηγό τους. Άρα λοιπόν, ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, να συζητήσουμε βεβαίως τους κανόνες λεπτομέρειές τους. Καθοριστική σημασία βέβαια είναι το πώς θα προχωρήσει η περαιτέρω να συζητησουμε βεβαίω του κανόνε λεπτομέρειε τους καθοριστικη σημασια βεβαια ειναι το πώ θα προχωρησει η περαιτερω επεξεργασια των δεδομένων και εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, παρασυρθεί το όλο εγχείρημα σε μια αδιαφανή ε, και ασαφή ζώνη στην οποία θα είναι σε θέση η, ε, ο κλάδος των αεροπορικών εταιριών να ελέγξει και να ξανακαλύψει όλα αυτά τα οποία εμείς προσπαθούμε να αποκαλύψουμε και άρα θα πρέπει να δούμε τι είδους ρόλο θα παίξει και ο σχετικός Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας τις αεροπορίες Γιατί υπάρχουν τρόποι να αποτραπεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανθρώπων που συνεργάζονται κανονικά και να ε, συγκαλυφθούν αυτές ε, οι πληροφορίες. Είμαι πάντως αισιόδοξη από τα άσκουσα από την συγκέντρια ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό συμπέρασμα, σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μερικές παρατηρήσεις μόνο και ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Τουβεγάκ. Πρόκειται για μια βασική νομίζω προϋπόθεση την εξασφάλιση ενός ε, ασφαλούς ενέργειου χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε, στο, να αξιοποιήσουμε στο μέσο τι δυνατότητε που θα έχουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια για το μέλλον. Βεβαίω θα πρέπει να, δίνεται, να γίνονται αυτέ οι αναφορέ περιστατικών, έστω και αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, Μεγάλη Βρετανία καταγράφει περισσότερε τέτοιε αναφορέ από ότι η Γερμανία. Οι τρόποι καταγραφής υπολογισμού των αριθμών αυτών είναι διαφορετικοί. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά πάντω έχει σημασία πάνω απ' όλα να γίνεται η αναφορά, να ε, καταγράφεται και να αξιολογείται στη συνέχεια, να αναλύεται. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει το προσωπικό εκείνο το οποίο θα έχει τη σχετική κατάρτιση για να μπορεί να αναλύσει τις πληροφορίες αυτές. Άρα λοιπόν με μια ενιαία ασφάλεια των μεταφορών, με ένα λειτουργικό, ε, με, με, με συλλογικούς θύλακες ε, ασφαλών, ε, ασφαλούς αέρια κυκλοφορίας, τι είδους ε, συνεργασία μπορούμε να περιμένουμε από τα κράτη-μέλη στον τομέα και της ασφάλισης βέβαια των πτήσεων και του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου πρέπει να προχωρήσει πολύ καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί όλα λένε δεν τα είναι. Και έτσι νομίζω μπαίνουμε λίγο πολύ και στο επόμενο θέμα της μεσης Ευχαριστώ, Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα γιατί καλύφθηκα σε πολλά από τα σημαντικότερα σημεία. Η συγγήτρια προφανώς ε, πολύ εύστοχα επισημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ε, προληπτικές ή προδραστικές όπως λέμε ε, δράσεις. Αυτό αποδεικνύουν οι πολλές αναλύσεις. Πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη λειτουργία της εναέρης κυκλοφορίας και βέβαια οι ελεγκτές εναέρειας ε, κυκλοφορίας και από την άλλη ίσως ο τρόπος με τον οποίο θα ε, παρακολουθούμε την αναφορά αυτών των περιστατικών αναπερίπτωση, τομέα κλάδο της ενέργειας κυκλοφορίας να πρέπει να διαφέρει. Αλλιώς θα συμπεριφερθούμε έναντι των μεγάλων αεροπορικών εταιριών και διαφορετικά σχέση με τις μικρότερες ιδιωτικές εταιρείες ιδιωτικής Σα Ευχαριστώ κύριο Κράμερ. Ε, ε, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Εδώ και δύο-τρία χρόνια είχα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ερώτηση όπου δεν έλαβα όμω ε, απάντηση για το δηλητηριώδε αέριο, για τον δηλητηριώδη ατμοσφαιρικό αέρα στην, στο σκάφο, μέσα στο αεροσκάφο fumes, όπως λέγονται ε, έχουν προκαλέσει δηλητηρίαση από την εισπνοή των αερίων αυτών σε πιλότους ε, αεροσκάφους τα αέρια αυτά. Πρέπει να σας πω ότι ακόμη και ο πρόεδρος του Bundestag που δεν είναι πολύ θετικά διακείμενος προς τους πρασίνους είπε ότι πρέπει πια να ε, ληφθούν μέτρα διότι Μπορεί να μην έχουμε ενιαίους ευρωπαϊκούς ουρανούς, αλλά έχουμε να κάνουμε με αεροσκάφη τα οποία κινούνται από το ένα κράτος στο άλλο και δεν μπορούν να, ε, να πούμε ότι περιορίζεται ο κίνδυνος που προξενούν ε, είτε στο ένα κράτος είτε στο άλλο. Κυκλοφορούν παντού, μας αφορούν όλους αυτά τα προβλήματα των δηλητηριωδών ε, αερίων στην καμπίνα του αεροπλάνου. Ε, δυστυχώς όμως δεν είναι δεσμευτική η καταγραφή των ε, περιστατικών. Ε, απλώς υπάρχει ένας κατάλογος, μάλλον ένα φυλάδιο το οποίο πρέπει θεωρητικά να συμπληρώσει ο αρμόδιος. Λέει περιστατικό ουδέν και ως εκ τούτου κλείνει η υπόθεση, δεν καταγράφεται δηλαδή. Άρα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά, χρειαζόμαστε αξιόπιστη κατάθεση αναφορά των περιστατικών συγκρίσιμη αναγνωσιμότητα και δεν είναι δυνατόν η Επιτροπή να σοπά και ο κύριος Κάλλας ιδιαίτερος, ε, γιατί ασφαλώς θα γνωρίσετε την ε, ερώτηση αυτή που έχω καταθέσει. Περιμένω λοιπόν από σας πλέον να αναλάβετε πρωτοβουλία. Δεν είναι δυνατόν, γιατί ξέρουμε ότι και κίνδυνο για σοβαρές ασθένειες αλλά και για θάνατο ακόμη μπορεί να αποδώσουμε στη, στα δηλητηριώδη αυτά αέρια μέσα στο αεροσκάφος. Ε, ξέρω ότι και πιλότοι σας έχουν αποστείλει επιστολές και έχουν αισθήσει την παρέμβασή σας. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πράτεται για αυτό ενώ αυτού μεγάλου κινδύνου και θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Ντεβιαγά και εντωμεταξύ αν είναι διτεθειμένη να ενσωματώσει στο κείμενό της ε, αυτά τα περιστατικά του δηλητηριώδους ε, ατμοσφαιρικού αέρα στην στα αεροσκάφη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κορνέλης, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έκανε καθώς το κείμενό της ορίζει ξεκάθαρα τα βασικά σημεία του κανονισμού και τις ε, κύριες προκλήσεις. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο σήμερα για τη συμβουλή του συζήτηση και το γεγονός ότι επεσήμαναν ε, αρκετά πολύ σημαντικά θέματα για το Ευρωκοινοβούλιο. Όπως ε, ανέφερε ιδίως η κυρία Φώστερ, ήδη υπάρχει νομοθεσία στον τομέα αυτό, μια οδηγία που εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια, οπότε δεν εφηρίσκουμε κάτι νέο. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε μια κείμενη πολιτική και καθώς θεωρούμε ότι η αναφορά περιστατικών είναι κρίσιμη σημασία στην όλη πολιτική, καθώς κινούμεθα ε, όλο και περισσότερο στην προσέγγιση με γνώμονα το κίνδυνο στην νομοθεσία μας. Θέλουμε δηλαδή βασικές πληροφορίες για το πού ελοχεύει ο κίνδυνος, οπότε η αναφορά περιστατικών είναι βασικό εργαλείο για να το επιτύχουμε αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σχεδόν όσοι πήραν το λόγο για αυτή τη συζήτηση ήταν θετικά αυτή την προσέγγιση. Ποιος είναι ο στόχος μας στην νομοθεσία. Όχι να, φεύρουμε, κάτι καινούργιο, αλλά να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε καλύτερα και να εδραιώσουμε την πολιτική επί συγκεκριμένων θεμάτων. Να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αυτά τα σημεία λοιπόν στα οποία θέλω να δώσουμε έμφαση είναι ακριβώ τα σημεία που και εσεί αναφέρατε στι παρεμβάσει Οπότε θα αναφερθώ εγώ μόνο σε τέσσερα θέματα. Πρώτα απ' όλα τίθεται το θέμα, ε, αν θέλετε, τη δικαιοσύνη που θα πρέπει να διέπει, Νοοτροπία μια δικαιοσύνη δηλαδή. Άρα θα πρέπει να προωθήσουμε μια τέτοια νοοτροπία αναφορά προσωπικών ακόμα και όταν ε, μιλάμε για ασφάλμα. Ε, που έχουν διαπραχθεί. Η πρόταση τη Κομισιόν περιέχει μια σειρά από νέε διατάξει με στόχο να προστατευτούν οι πάλι στην ε, αεροπορία από τη Μόρια, ώστε να μπορούμε να ενθαρρύνουμε την αναφορά προστατικών, χωρί αυτό να του δίνει πλήρη ασυλία όταν ε, μιλάμε για την περίπτωση βαριά αμέλεια, ιδίω η πρόταση προστατεύει όσου κάνουν αυτήν την αφορά από προκατάληψη ή από ψόχο από τον εργοδότη. Επίσης διασφαλίζει η πρότασή μας ότι όλες οι οργανώσεις ε, θα υιοθετήσουν ε, ένα εσωτερικό κανονισμό, αν θέλετε, διοντολογία που να βασίζεται στη δικαιοσύνη και είναι ένα σημείο το οποίο ανέφεραν όλοι όσοι πήραν το λόγο στη συζήτηση και είναι, αν θέλετε, από τις πλέον δύσκολες ε, συζητήσεις που αυτή τη στιγμή έχουμε ανοιχτές με τα κράτη-μέλη επί της πρότασης, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικές νοοτροπίες σε ό,τι αφορά το ποινικό και το αστικό δίκαιο. Οπότε πραγματικά είναι ένα από τα πλέον ε, δύσκολα σημεία του κανονισμού που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεύτερο και βασικό στοιχείο σε αυτό το κανονισμό είναι να θεσπίσουμε μηχανισμού τέτοιους ώστε τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται και καταγράφονται να μπορούν να χρησιμοποιούνται τον καλύτερο τρόπο. Οπότε ε, έχουμε νέε υποχρεώσει για την ανάλυση των πληροφοριών ασφαλεία που συλλέγονται και να εντοπίσουμε και να κάνουμε ένα follow-up για τα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για να αντιμετωπίζονται ε, τυχόν ελλείψει. Απαιτήσει που δεν ε, είναι παρούσε στην κείμενο οδηγία και γι' αυτό θεωρούμε ότι το σύστημα έω τώρα δεν είναι πλήρω αποτελεσματικό με βάση το κείμενο νομικό πλέον πλαίσιο. Τρίτον, η πρότασή μας προωθεί μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την ΕΑΣΑ. Σήμερα η ανταλλαγή πληροφοριών δεν ε, γίνονται πλήρω σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίω αφορά προστατικά στον αέριο χώρο ε, μια χώρα ε, και ενημερώνεται ε, το τυχόν ενδιαφερόμενο κρατός μέλος. Η ΆΣΕ, για παράδειγμα, δεν ενημερώνει για α, θέματα που, που συμβαίνουν στον ένα χώρο το οποίο είναι υπεύθυνοι. Όπως ανέφεραν πολύ εκτός Κοινοβουλίου, ο ρόλος της ΕΑΣΑΝ προκειμένου είναι κρίσιμη σημασία για την αναφορά περιστατικών και θέλω να σας καθησυχάσω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα σε αυτόν τον κανονισμό και ε, τους υφιστάμενους τεχνικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς όπως ο 216 του 2018 καθώς εκεί υπάρχουν τις ε, απαιτήσει αναφοράς περιστατικών, αλλά αφορούν πολύ συγκεκριμένα τον χώρο που λαμβάνουν τα περιστατικά. Είναι συμπληρωματικές λοιπόν αυτές οι διατάξεις και δεν έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Στόχος είναι να, έχουμε τελικά ένα οριζόντιο καθολικό σύστημα που να βοηθήσει την καλύτερη εφαρμογή της ε, οδηγίας. Επίσης, στην πρότασή μας δίνουμε στην ΕΑΣΑ πολύ πιο κεντρικό ρόλο στο όλο σύστημα, δίνοντας πρόσβαση στην υπηρεσία σε όλες τις εκθέσεις, όλες τις αναφορές μέσω μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, έπειτα δίνουμε στην ΕΑΣΑ τον ρόλο της ανάλυσης όλων αυτών των στοιχείων και την, το καθήκον του follow-up και όλα τα θέματα που αφορούν την πιστοποίηση και το αξιόπλο των αεροσκαφών είναι στοιχεία που διαβιβάζονται άμεσα στην ΕΑΣΑ. Και θέλω να πω ότι είναι στοιχεία θα συλλέγονται λοιπόν στην κολονία και ε, θα τα συλλέγει και θα τα επεξεργάσει τη γραμματεία της ΕΑΣΑ. Τέταρτο και τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω στην πρότασή μας είναι ότι η πρόταση αναφέρει ότι πέρα από το αναγκαίο έργο που πρέπει να γίνει σε δανεικό επίπεδο από τη βιομηχανία και τα κρατημέλη, το δίκτυο αυτό που σας ανέφερα θα συσταθεί επισήμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αποτελείται από τον προγνώμονα των κρατών μελών και το συντονισμό θα έχει η ΕΑΣΑ. Ε, με στόχο την ασφάλεια μέσω της αναφοράς ε, σημαντικών περιστατικών που μπορούν να μας υποδείξουν κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές που υπάρχουν και μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτό το επίπεδο. Είμαστε ε, απόλυτα πεπισμένοι ότι με αυτή την πρόταση θα αποφύγουμε σημαντικά ατυχήματα σε αερομεταφορές και θα μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ίσως ακόμη ένα σχόλιο να κάνω το οποίο δεν έθιξα πέρα από τα βασικά σημεία που ανέφεραν ε, οι συναδελφοί σας και αφορούν το ρόλο της ΕΑΣΑ. Πολλοί ε, αναφέρθηκαν στην γενική αεροπλοεία και ε, στα ελαφρά αεροσκάφη και από ό,τι κατάλαβα θέλετε να καλυφθούν και αυτές οι κατηγορίες από αυτό το κανονισμό. Συμφωνούμε και εμείς καθώς λοιπόν κινούμεθα σε μια σειρά προς μια σειρά ρυθμίσεων που θα είναι, είναι λιγότερο επιλεστική, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερα καθήκοντα και πιο σημαντικό ρόλο στους ίδιους τους υπαλλήλους, στους πιλότους ε, και το πλήρωμα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη πρωτοβουλία οι εργαζόμενοι, αλλά αναλογικά, καθώς ε, τα λεφτά σκάφη δεν είναι το ίδιο πράγμα όπως ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος και επίσης η συχνότητα και το είδος των περιστατικών θα πρέπει προκειμένου να προσαρμοστούν. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα βασικά σημεία και ευχαριστώ πολύ. Thank you. I don't think you are... Ευχαριστώ. Δεν απαντήσατε στον κύριο Κράμερ όμως, κύριε Κορνέλισον. Θα το κάνετε κάποια στιγμή. Τώρα, ναι. Ναι, συγγνώμη, πρόεδρε για το θέμα της ποιότητας του αέρα μέσα στην καμπίνα πιβατών. Θα σας στείλουμε και γραπτά πλήρη απάντηση, αλλά τι θα λέει. Θα λέει ότι η Άσα εξετάζει αυτό το θέμα, το έχει εξετάσει, έχουν μελετήσει το θέμα, έχουν ε, προβεί και σε μετρήσεις μάλιστα μέσα ε, στα αεροσκάφη δεν ε, όμως έχουν καταλήξει πραγματικά σε συμπεράσματα, οπότε δεν αναλαμβάνεται καμία δράση επί του παρόντος, γιατί δεν είναι καταληκτικά τα δεδομένα τα οποία συνέλεξαν, ώστε να μπορούν να καταλήξουν και στο τι πρέπει να γίνει. Όσο περισσότερα στοιχεία πάντως προκύπτουν, η Άζα τα εξετάζει. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα σε ορισμένες χώρες, μέλη μάλιστα, που δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Πάντως το θέμα αυτό, της ποιότητας δηλαδή το αέρα μέσα στο ροσκάφος, θα καλύπτεται από τον υποχρεωτικό κατάλογο περιστατικών που θα πρέπει να αναφέρονται. Και να λοιπόν ένα καλό παράδειγμα μια περίπτωση δηλαδή που θα προχωράει μετά και στο καθορισμό πολιτικής ανάλογα. Κύριε Κράμερ, βλέπω θέλετε. Καλά, γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μα δεν είναι μεμονωμένου κράτους μέλους το πρόβλημα. Απλώς σε κάποια κράτη-μέλη αποφασιστικά γίνονται έρευνε, ενώ σε κάποια άλλη συγκαλύπτεται και λένε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και, πρέπει, και εσεί από την άλλη περιμένετε να προκύψει δυστύχημα για να αποφασίσετε να αναλάβετε δράση. Τρία χρόνια έχουμε αυτή την υπόθεση αυτή. Όποιο ε, κυβερνήτη αεροσκάφου καταγγείλει τέτοια περιστατικά κινδυνεύει από διακριτική μεταχείριση και δεν τολμάει να κάνει τέτοια δήλωση, διότι φοβάται τέτοια αναφορά, διότι φοβάται ότι θα χάσει τη θέση του. Τι κάνετε, περιμένετε να γίνει δυστύχημα, σα το λέω ξεκάθαρα, θα είσαστε συνυπεύθυνο. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Κράμερ. Όχι. Καλώς. Να ξεκαθαρίσω όμως τι λέτε κύριε Καρνέλης. Να λέτε ότι η ποιότητα ε, του αέρα θα καλύπτεται από τον κατάλογο. Έτσι, κύριε Ντεβεράκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να ακούσω τα πρώτα σχόλια που έχετε για το θέμα αυτό και βλέπω ότι συμφωνούμε και όλοι θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική έκθεση αυτή. Στο πεδίο εφαρμογή φυσικά και πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Πρέπει να ισχύει για όλη την αεροπορία. Βέβαια δεν μπορεί να υπάρχουν ίδιοι κανόνες για τα μικρά και τα μεγάλα αεροσκάφη. Όσον αφορά τώρα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροπορίας, την ΕΑΣΑ, εννοείται ότι δεν θέλουμε να αποκλείσουμε τον οργανισμό αυτό κάθε άλλο, γιατί είναι τεράστια σημασία και πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο στην ανάλυση των περιστατικών που αναφέρονται. Συμφωνούμε για το ότι θέλουμε όσο γίνεται περισσότερη προστασία για αυτούς που αναφέρουν περιστατικά. Αν ε, οι πιλότοι ξέρουν ότι προστατεύονται, ε, τότε θα αναφέρουν περισσότερα περιστατικά εφόσον υπάρχουν. Και αυτό προσπαθεί να κάνει το κείμενό μου, να υπάρχει αυτή η νοοτροπία της δικαιοσύνης. Όπως είπε και ο κύριος Κιούν, πρέπει να φροντίσουμε πάση θυσία να γίνεται στη συνέχεια καλή ανάλυση δεδομένων. Τώρα για το περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε κύριε Κράμερ, είναι οι πυρογνώμονε οι οποίοι θα αποφασίσουν κατά πόσο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο ή όχι. Πάντω είναι από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπουν στον κατάλογο και όχι στο κυρίω σώμα του κανονισμού. Ο κατάλογο θα είναι παράρτημα στον κανονισμό. Λοιπόν, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να έχει μια ισχυρή θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα για να ενισχυθεί η ασφάλεια στην αεροπορία. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. σε ευχαριστώ πολύ. να ξέρετε ότι στις 17 Ιουνίου θα παρουσιαστεί η έκθεση, τότε θα καθοριστεί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που θα είναι 27 Ιουνίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 17 Σεπτεμβρίου και θα πάει το θέμα στην Ολομέλη Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, 17 Ιουνίου θα έχουμε την έκθεση, προθεσμία για καταθέση τροπολογιών θα είναι 27 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 17 Σεπτεμβρίου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέβερακ. Και το επόμενο θέμα είναι τα αέρια του θερμοκηπίου με εισηγητή τον κύριο Μπαρνιό που είναι επί της ουσίας αρμόδια για την έκθεση αυτή η Επιτροπή Περιβάλλοντος και ο κύριος Αλκαντράουι και άλλοι είναι εδώ. Ωραία. Κύριε Παρνιό, ξεκινήστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παρνιό δεν μπορεί να είναι σήμερα, λέει ο κύριος Αλκαντράουι που τον αντικαθιστά. Έπρεπε να είναι στο εξωτερικό, οπότε θα σας παρουσιάσω εγώ τις κύριες γραμμές της, γνωμο... της γνωμοδότησής του αυτής. Ξέρετε ότι τα αέρια αυτά του θερμοκηπίου επιβάλλουν μια αλλαγή στο κλίμα και ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ πιο επιβλαβή από άλλα αέρια του θερμοκηπίου. Εμείς θέλουμε μια οικονομία ανταγωνιστική που να έχει βέβαια χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όμως οι εκπομπές άλλων αερίων του θερμοκηπίου, των ε, φθοριούχων αερίων ε, κτλ πρέπει να μειωθούν 72-73% μέχρι το 2030. και 78% μέχρι το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στα τέλη του 2012 υιοθέτησε τον κανονισμό αυτό και διάφορα μέτρα όσον αφορά την επεξεργασία που γίνεται στα φθοριούχα αυτά αέρια στο τέλος της ζωής τους. Ο κανονισμός αυτός τώρα προβλέπει τη μείωση διάθεσης στην αγορά φθοριούχων αερίων που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με μέσω ποσοστώσεων και με επιπλέον απαγορεύσεις όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμών ή μηχανημάτων τα οποία περιλαμβάνουν φθοριούχα αέρια που επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όσον αφορά τώρα τις μεταφορές. Προτείνεται από την Επιτροπή αλλαγή του πεδίου εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού επεκτείνοντας τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την επεξεργασία. Είτε πρόκειται για την πρόληψη των εκπομπών, είτε πρόκειται για τον έλεγχο της μόνωσης, είτε πρόκειται για τις διαρροές, είτε πρόκειται για ένα μητρό που καταγράφονται τα αέρια αυτά, αλλά περιλαμβάνει και την φόρτωση των φορτηγών ψυγείων. Μιλάει για τη μείωση της διάθεσης στην αγορά των ε, HFC 134, HFC 125 και HFC 143 που είναι οι κλωροφθοράθρακες είτε πρόκειται για μείγματα είτε πρόκειται για την καθαρή τους μορφή καθώς και την απαγόρευση των λόγω σκοπούς εξυπηρέτησης και συντήρησης. Τώρα, στο ψήφισμά του 14 Σεπτεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για την ταχεία σταδική κατάργηση της παραγωγής και της κατανάλωσης υδροχλωροφθοροανθράκων σε διάφορα προϊόντα και εφαρμογές. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν ανταποκρίνεται στο στόχο αυτό, αλλά ο πιστεύει πιστεύει το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να διευρυνθεί περισσότερο, προσέχοντας όλος ιδιαίτερος στο θέμα της κοπιμότητας. Όσον αφορά τους ελέγχους για διαρροές, η πρόταση καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος των μεταφορών, και εστιάζεται αποκλειστικά στα φορτικά ψυγεία άνω των 3,5 τόνων και στα ρημουλκούμενα ψυγεία. Ο συντάκτη λοιπόν εκτιμώ ότι δεν είναι σκόπιμο αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογή των φορτικών ψυγείων κάτω των 3,5 τόνων, των ημιφορτικών ψυγείων και των εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων λόγω του αριθμού οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων που κυκλοφορούν στην Ένωση. Επιπλέον, το πεδίο αυτό εφαρμογή το περιορισμένο θα μπορούσε να δημιουργήσει και διακρίσει εντό του ίδιου του τομέα. Στην έκθεση αυτή ο Ζήλ υπενθυμίζει ότι οι τομεί των συνδρομικών και των θελασσιών μεταφορών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου. Ωστόσο, ο τομέα των θελασσιών μεταφορών, λόγω τη ιδιωτερότητέ του και κυρίω του διεθνού χαρακτήρα του, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδική νομοθεσία, όπω προτείνει η Επιτροπή. Φυσικά και θέλουμε το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού να επεκταθεί όσον αφορά τον έλεγχο τη ε, διαρροή ο περιορισμός όμως της παραγωγής των αερίων αυτών για την ε, συντήρηση μετά το 2020 δεν πρέπει να εφαρμόσετε στις μεταφορέ γιατί το κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο, θα δημιουργούσε υπέρμετρο κόστος, δηλαδή για τις επιχειρήσεις που θα υποχρεώνονται να αντικαταστήσουν, να τροποποιήσουν τον εξοπλισμό τους πριν από το τέλος του κύκλου ζωής, χωρίς να εξασφαλίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη άλλα μέτρα ε, φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά καλά προσαρμοσμένα στη μεταφορά, όπως είναι η εκ των προτέρων γόμος, η τήρηση μητρών. Όσον αφορά τώρα τον εφοδιασμό με εναλλακτικά αέρια. Ο τομέας των μεταφορών το 2012 έλεγε ότι υπάρχουν προβλήματα για ορισμένα αέρια και θέλουν να καθυστερήσει η οδηγία ΚΜΟ. Τα φθοριούχα αέρια με χαμηλότερο δυναμικό πλανητικής αύξησης θερμοκρασίας, που εξετάζονται ως βραχυπρόθεσμη μεσοπρόθεσμη λύση, βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ακόμα. Συνεπώς, ο Ζήλ προτείνει να είναι χαλαρότερο το χρονοδιάγραμμα για τα πρώτα έτη εφαρμογή και ζητεί και αξιολόγηση του κανονισμού μετά το πέρας τη περίοδου αυτής, προκειμένου να υπάρξει αναπροσαρμογή του χρονοδιάγραμματος αν χρειάζεται. Εν κατακλείδη, υπογραμμίζω τα θέματα ασφαλεία των αλλακτικών αερίων καθώς και οι ενεργειακές τους επιδόσεις πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Ορισμένα εναλλακτικά αέρια είναι έφλεκτα και ενδέχεται να παρουσιάζουν πρόσθετους κινδύνους σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Όσον αφορά τις ενεργειακές αποδόσεις, θα πρέπει επίσης να είναι ισοδύναμες τουλάχιστον των αερίων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ώστε να μην προκαλούν εκπομπές διοξιδίου άνθρακο εξαιτία της αυξημένης τελικά κατανάλωση των οχημάτων. Υπενθυμίζω επίση ότι η ημερομηνία 26 Απριλίου είναι προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Στι 29 Μαου θα εξεταστεί στην Επιτροπή μα η έκθεση αυτή και 30 Μαου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μα. Κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβριο θα πάει έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλκαδράουι. για την τόσο ωραία παρουσίαση για το ΕΛΚΑ. Κύριε Σπάνης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο. Αυτό το σχέδιο κανονισμού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση της ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η Επιτροπή ουσιαστικά μας διατυπώνει μέτρα και προτάσεις που γίνονται σωστή κατεύθυνση. Βασική συζήτηση, εν προκειμένου, αφορά πώς μπορούμε να ε, κινηθούμε ταχύτερα και τι περιορισμούς θα πρέπει να θέσουμε έως το 2020. Τομείς ε, μπορούμε να λάβουμε δράση και όπου δεν έχουν οριμάσει συνθήκε για τέτοια επιτάχυνση δικασιών. Δεν έχουμε τέτοια πρόοδο στον τομέα της καινοτομία ώστε να μπορέσουμε να εξέφερουμε αυτά τα εναλλακτικά αέρια. Επίσης, τα ποσοστά επιπλαβών ρήπων δεν δικαιολογούν μια τέτοια ε, προώρη εισαγωγή των λακτικών αερίων. Και αν με επιτρέπετε, θέλω να αφαιρθώ σε αυτούς τους τρεις ε, τομείς που δείξατε και στην παρουσίασή σας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά μικρού μεγέθους. Είπατε και συμφωνώ ότι η προθεσμία εισαγωγή του 2020 δεν είναι ρεαλιστική ο στόχο. Αυτό που μπορούμε να προσδοκούμε είναι ότι θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, ώστε να μας ε, δοθεί η δυνατότητα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να βρούμε εναλλακτικές λύσεις ε, που δεν ε, θα θέσουν σε κίνδυνο το στόχο του 2020. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στις βιομηχανικές τεχνικές ψήξεις. Η κύρια Επιτροπή έχει εκφράσει ανησυχίες επ' αυτού, γιατί στο αρχικό της paper πρόβλεπε νωρίτερη καταλεκτική προθεσμία, μετά αναθεώρησε, γιατί και η ίδια η Κομισιόν δεν θεωρούσε πλέον εφικτή αυτή την προθεσμία του 2020, δηλαδή να εισαχθούν τέτοιε νέε τεχνικές έω τότε. Βεβαίω, η μηχανή τροφίμων ήδη υπάρχουν τέτοιου, τέτοιες κατηγορίες κλιματιστικά και θα μπορούσαν λοιπόν να τηρήσουν με το 2020. Σε ό,τι αφορά την, ε, τους μηχανισμούς ψήξης ε, στα μεταφορικά οχήματα, όταν κινούμαστε στα περιβάλλοντα κάτω των 50 βαθμών Κελσίου, εκεί πιστεύω τα εναλλακτικά αέρια δεν είναι διαθέσιμα ακόμη. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές τεχνικές ψήξεις, έχει επιτευχθεί πρόσφατα ε, αξιοθαύμαστη πρόοδος, αλλά να μην ξεχνάμε κάποιες ιδιαίτερε συνθήκες ε, και γεγονότα στη Μεσόγειο, όπου κάποιοι έμποροι έχουν αγοράσει πρόσφατα μηχανισμούς ψήξης που σύντομα θα απαγορευθούν λόγω ε, των αερίων που εκπέμπουν. Αυτό ε, συνεπάγεται σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων και θα ε, υπονομεύσει σημαντικά την αντιγωνιστικότητά τους. Αν δεκαπλασιαστεί συζητούν οι επιλέξιμες κατηγορίες, αυτό μπορεί να διευκολύνει τους μικρούς εμπόρους, όχι όμως τους μεγαλύτερους. Σε αυτούς το τομείς χρειάζεται να γίνει περαιτέρω δουλειά. Ε, και από αυτό έχω κάνει και κάποιες προτάσεις. Yeah, vielen Dank. Η κυρία Μάχινερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Πανιά, ο οποίος έκανε την επεξεργασία του θέματος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, αέρια τα οποία μπορεί να έχουν μόνο 2% από το ποσοστό των αερίων θερμοκηπίου αυτή τη εποχή, αλλά έχουν ανωδική τάση και ως εκ τούτου πολύ σωστά δεδομένων και των προσπαθειών για περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα να έχουμε και μία πρόταση για το θέμα αυτό. Για τα οχήματα λοιπόν, τον τομέα των μεταφορών ειδικότερα, έχουμε να κάνουμε με ε, εγκαταστάσεις γόμωσης ή ψήξης αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τα οδικά οχήματα, τα οχήματα για χρήση στους δρόμους, αλλά και στους σιδηροδρόμους, σιδηροδρομικές μεταφορές, τελευταίες μεταφορές κτλ. Και θα πρέπει οπωσδήποτε όταν είναι και επικίνδυνα αυτά αερία να τα αντικαταστήσουμε με κάποια εναλλακτικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει και πολύ σωστά επισημαίνει και ο ή ο κύριος Ελκαντράου εκ μέρους του, ή ο συνάδελφος από το ΕΛΚ, ε, να αξιολογηθεί το πόσο εφικτά, εφικτό είναι να χρησιμοποιηθούν τα αναλλακτικά αυτά αέρια. Όταν λοιπόν λέμε για κάποιο αέριο ότι θα πρέπει να, να αντικατασταθεί, να απαγορευτεί, θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικά στοιχεία με συγκεκριμένη εστίαση στις στρατηγικές μας, αν τις εξυπηρετεί δηλαδή η εναλλακτική λύση, χωρίς να φέρνει πλέον προβλήματα ή κινδύνους. Ο κύριος Συγητής προτείνει κάθε πέντε χρόνια να γίνεται μια αναφορά, ε, καταγραφή, πολύ καλή πρόταση, διότι αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το περιβάλλον ε, ή την ασφάλεια, καλό θα είναι να μπορούμε να παρακολουθούμε ανά πενταετία την κατάσταση. Και επίσης, όπως και οι συνάδελφοι που μίλησαν νωρίτερα, πιστεύω ότι θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε τα εναλλακτικά αέρια. Ως προς τις εκπομπές θα πρέπει να βρούμε μια λογική λύση και βεβαίως ε, ο κύριος Γκρός με την ε, έκθεση του για τη Λευκή Βίβλο έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Κύριε Τέιλορ, μόλις ήρθατε, θέλετε να πάρετε μια ανάσα ή είναι η σειρά σας τώρα. Έχετε το λόγο. Yes, it's well. It's the sun is not yet uh, over the yard arm, as they say. Oh, thank you very much, Chair. Uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη και λυπούμε τα που έχασα το μεγαλύτερο κομμάτι της συζήτησης, αλλά με χαρά δράτω με τις ευκαιρίες να τοποθετηθώ πολύ σύντομα για την έκθεση. Για τα αέρια F και το σχετικό κανονισμό. Ε, με απασχόλησε το γιατί έφτασε στην Επιτροπή των Μεταφορών το θέμα αυτό. Μέχρι ότου κατάλαβα ότι έχουμε γομωμένα ε, ε, φορτηγά και αντίστοιχα άλλα οχήματα και ως εκ τούτου σημαντικό είναι για την Επιτροπή των Μεταφορών ο εξοπλισμός, η τα μηχανήματα στα οποία εστιάζονται αυτά, ε, ε, βρίσκονται εκτοποθετημένα αυτά τα αέρια, να ε, είναι ασφαλής ύστερα από μία πρόσκρουση, από ένα χτύπημα στο δρόμο, υπάρχει κίνδυνος της διαρροής. Οι τροπολογίες λοιπόν του κυρίου Παρνιού ενδέχεται ωστόσο να οδηγήσουν σε υπερβολικά δεσμευτικές λύσεις ως προς τη σταδιακή εξάλληψη. Μάλλον του κυρίου Άικχαουτ και του κυρίου Λάινεν από την Επιτροπή των Μεταφορών ε, τις προτάσεις θα προτιμήσω, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ πιο κοντά στο πρότυπο της Επιτροπής και όπως είπα, ε, μέχρι τις προτάσεις του κύριου Άικαουτ και του κύριου Λάινεν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι υπερβολική η δέσμευση. Για το αν θα πρέπει να προχωρήσουμε στις, μετα... στις απαγορεύσεις του τομέα των μεταφορών. με στόχο να περιορίσουμε το δυναμικό υπερθέρμανσης, πλανητικής υπερθέρμανσης των αερίων που χρησιμοποιούνται. θα πρέπει στο, στην ψήξη να ζητήσουμε την απαγόρευση των ε, χειρότερων ε, τύπων υδροχλωροφθορανθράκων από τα ψυγεία, φορτηγά ψυγεία κυριμικούμενα. Όσον αφορά τις ε, μεταφορές επιβατών μέχρι το 2027, τα λεωφορεία μέχρι το 2020, ε, λίγο πολύ αυτά είχαν από πρόεδρε και πρέπει να ακούσω και ότι προλάβω από τη συζήτηση και να δω και τις τροπολογίες. Κύριος Ζήλας, Ζήλε, θέλετε και εσείς να πιείτε μια γουλίτσα. Ναι, εμείς από το ECR εν γέννη υποστηρίζουμε τις πιο περιβαλλοντικές και οικολογικές λύσεις σε σχέση με τα αέρια τύπου F. Αλλά πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε για τις επιπτώσεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση και την επιτάχυνση αυτής, εμείς είμαστε κατά κάθε λύση που θα επιτάχυνε την κατάργηση σε σχέση με τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν επαρκείς ποσότητες των αναλλακτικών ε, εγκαίρος. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την επιστολή ευελιξία που προτείνει ο εισηγητής. σε σχέση με την ε, διάθεση υδροχλωροφθορών στην αγορά ως προϋπόθεση. Η κατάργηση εξοπλισμού με δυναμικό γόμος μέχρι τους 5 τόνους πάλι θα έχει κίνδυνο για επιβάρυνση γραφειοκρατική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την χρήση σε οχήματα ε, φορτηγά και φορτηγάκια με 3,5 ε, τόνους πάλι έχουμε ανησυχίες. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται δηλαδή ε, περιτά με κόστος αφόρητο και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο τομέας των μεταφορών. Το θέμα της κατευσούδωτης συμπράξεως είναι άλλο ζήτημα. Στο παράρτημα 5 έχουμε ποσοστώσεις για τους υδροχλωροφθορανθρακές και προτείνουμε τις ποσότητες αυτές να τις καταγράψουμε στο άρθρο 19. Ευχαριστώ, Φώστρο. Yeah, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζήλερ κάλυψε πολλά από αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Αλλά έχω μερικά επιπλέον ε, σημεία να προσθέσω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Γιατί είτε πρόκειται για τέσσερις τόνους λαχανάκια είτε δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, αλλά μερικές φορές τα ψυγεία αυτά μεταφέρουν φάρμακα. Ό,τι και να γίνει στο μέλλον δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει αναλλακτική λύση και όχι να αναπλώσει ευσεβή σπόθη. Όσον αφορά τώρα τα ρευματοκιβώτια, τα containers, δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να τα συμπεριλάβουμε. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προφανώς θα έχει άλλη άποψη. Έπειτα υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Για τη συντροπολογία 6 μιλάμε για 5 χρόνια, ενώ στην 5 για 11 χρόνια. Είναι αντιφατικά μεταξύ τους πέντε χρόνια για μας είναι πολύ λίγο. Αυτά που πάνε οι συνάδελφοι πάντως με έχουν καλύψει και συμφωνώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος ε, Ρίπκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, ανάμεσα στα θωριούχα αέρια και τους χλωροφθοράνθρακες που είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στα ροζόλ και έχουν απαγορευτεί. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ τους. Ποια ακριβώ είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες θωριούχων αερίων. Έπειτα οι μεταφορές όσον αφορά την χρήση τέτοιων αερίων πόσο παρεμβαίνουν με τα ψυγεία, για παράδειγμα τα φορτικά ψυγεία κλπ. Και τρίτη και τελευταία μου ερώτηση. Ο κλιματισμός των ΙΟΤΑΧΗ αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό τέτοιων ε, φθοριούχων αερίων. Πολύ σύντομα. Γιατί σε σχέση με τα ιδιωτικά, ιδιωτικής χρυσού αυτοκίνητα. Θα θέλω να το διετύπωση το κυρία Ρικέ. Ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να ρωτήσω εάν έχει υπολογίσει το συνολικό κόστος από την εισαγωγή αυτών των μέτρων. Διότι άλλος λέει ότι μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά κάποια κατηγορία μεταφορέων. Άλλοι λένε όχι. Πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία. Γιατί τι εναλλακτικέ τα εναλλακτικά αέρια που προτείνονται θεωρούνται όλα ασφαλή. Διότι γίνονται πολλά ερωτήματα και ως προς την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία και επειδή από την εμπειρία που έχουμε από την νομοθεσία με τη σχετική με τις ε, ενώσεις, τεχνολογικές ενώσεις, ε, βλέπω ότι τείνουμε να εισάγουμε λύσεις οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί απολύτως και που τελευταία στιγμή χρειάζεται να τροποποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η Επιτροπή να μας εξηγήσει με βάση και τις προθεσμίες που προτείνει πόσο βέβαια είναι για το εφικτό της εισαγωγής αυτής της διαφορετικής τεχνολογίας. Είναι ένα θέμα δύσκολο και ποιος διαβάσει αναφορές τεχνικών, ειδικών, που είναι μεταξύ τους και πολλές φορές ε, αμφιλεγόμενες και αντικρουόμενες, είναι πολύ δύσκολο να ε, πει κανείς με ευκολία ότι μπορεί να προτείνει την τάδε λύση και έτσι ως εκ τούτου ένα καλό νομοθέτημα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει πολύ να σπροσκεφαλιάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πριν ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο, θα ήθελα και εγώ, όπω και άλλοι συνάδελφοι, να υπογραμμίσω ότι το θέμα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στις μεταφορές, έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Από τη δική μου εκλογική περιφέρεια ξέρω πολύ καλά ότι ιδιαίτερα οι ασθηματικοί χρησιμοποιούν σε ε, σπρέι που εισπνέουν για την αντιμετώπιση του άσθηματος τέτοιου είδους αέρια. Άρα υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό θα θέλαμε να δούμε μια πλήρη ανάλυση συνεπειών και αποτελέσματος. Κύριος Ρέιναρ, από τη Γενική Διεύθυνση για την Κλιματική Αλλαγή. Πού είσαστε. Περάστε. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. So we got a number of very precise... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα και θέλετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα ήθελα βεβαίω και εγώ να παραπέμψω στη μελέτη αντικτύπου την οποία κάναμε και σας παρουσιάσαμε με βάση μια εμπεριστατωμένη πραγματικά μελέτη του όλου τομέα η οποία μελέτη δίνει ακριβείς απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τομεακά αναλύοντας και τις διαθέσιμες εναλλακτικές ε, λύσεις και το δυναμικό απορρόφησης αυτών από την αγορά στο μέλλον. Με τη μεγάλη δικτύπου και την πρότασή μας, ακολουθήσαμε πρώτα απ' όλα μια πολύ στρατική προσέγγιση. Δεν ε, εξετάσαμε καθόλου εναλλακτική τεχνικές λύσεις που να είναι πλήρως διαθέσιμες και που να είναι α, εξίσου ασφαλείς όπως οι υδροχλωροφθοράνθρακες. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κριτήρια αποκλεισμού εναλλακτικών αερίων. Και καταλήξαμε λοιπόν κάποια στιγμή στο συμπέρασμα ότι όταν έχουμε μικρά κινητά κλιματιστικά, τα οποία ε, μπορεί να απαγορευτούν με την πρότασή μας, αυτό το κάναμε καθώς είχαμε ένα θετικό συμπέρασμα ότι ήδη υπάρχουν εναλλακτικά ε, αέρια των, των ε, Υπάρχουν λοιπόν εναλλακτικά αέρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Ετέθη ένα ερώτημα. Υπάρχουν ε, εναλλακτικά αέρια αποστασίευσης που χρησιμοποιούνται στα σπρέι και ε, ποια θα είναι η διαφορά σε σχέση με αυτά τα αέρια που χρησιμοποιούνται σήμερα. Ναι, υπάρχουν και εναλλακτικά αέρια των υδροχλωροθρανθράκων, αλλά έχουν αντικατασταθεί από μη ε, υδροχλωρούσες ε, τέτοιες ουσίες. Σχετικά με την κατάσταση στην αγορά και το μερίδιο της αγοράς θα εξηγούμε εξελικτικά τα αεροζόλ ως μελτίου της αγοράς είναι κάτι κάτω από 10% του συνολικής χρήσης, ενώ η ψήξη είναι περίπου το 80% της χρήσης αυτών των αερίων. Άρα είναι ο κύριος ε, τομέας χρήσης αυτών των αερίων, η ψήξη. Γενικά, βλέπουμε πολύ θετικά την γνωμοδότησή σα και το γεγονός ότι η γνωμοδότησή σα συμφωνεί με τη γενική προσέγγιση που ακολουθήσαμε. Όμως, με τη συντηρητική αυτή προσέγγιση που εμείς επιλέξαμε για αυτό το πέρασμα ε, στη νέα, στα νέα αέρια, η επιβράδυνση της όλης διαδικασίας θεωρούμε ότι θα μας ε, οδηγεί στο να χάσουμε κάποιες ευκαιρίες. Υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε με τους ρυθμούς που εμείς προτείνουμε τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό ε, και τώρα αναφέρουμε στο τομέα των μεταφορών συγκεκριμένα, πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε τον ε, ισότιμο ανταγωνισμό σε όλους τους τομείς των μεταφορών. Γιατί δεν συμπεριλάβουμε τα κοντέινερ, για παράδειγμα, λόγω των ησυχιών τρέφουμε για την εφαρμογή αυτών των μέτρων που αφορούν τον εξοπλισμό των κοντέινερ που θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Αναφέρομαι ιδίως στα πεμπτοκιβώτια που κινούνται και με τις θαλάσσιες μεταφορές. Κατά πόσο λεπτό δηλαδή θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο στην πρότασή μας είναι η απαγόρευση στην ε, γόμωση του υλικού. Ένα μέτρο που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και τέτοιο εξοπλισμό που, περιέχει, που ε, έχει γίνει γόμωση των αερίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Βεβαίως ε, μπορούν να παρακάμψουν τον κίνδυνο με την εισαγωγή αυτού του εξοπλισμού, αυτών των προϊόντων στην Ένωση. Γι' αυτό κρατήσαμε και πολύ ανοιχτό το πεδίο εφαρμογή. Αν ε, απαιτείται περαιτέρω ευθυγράμμιση και συντονισμό για να αντιμετωπίσουμε ειδικά την περίπτωση των μέσων μεταφορά, είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε. Επίσης, η απαγόρευση ε, στην χρήση πολύ ε, υψηλών σε περιεκτικότητα Ε, Ναι, εμείς προτείνουμε ε, τους πεντατόνους. Αυτό το μέτρο δεν έχει σκοπό να εξαναγκάσει τους εμπόρους στην αντικατάσταση του εξοπλισμού. Αφορά μόνο τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να γίνει αλλαγή του μηχανισμού ψήξης χωρίς να γίνει πλήρης αντικατάσταση του συστήματος. Και εδώ, αν ζητήσετε κάποια τροποποίηση, ε, επιμέρους τροποποίηση του πεδίου εφαρμογή, να μπορούμε να εξετάσουμε κάποια επιχειρήματα, καθώς είναι κάτι που έχουμε λάβει υπόψη και το έχουμε δει και σε κάποιες τροπολογίες σας ε, έως τώρα. Έπειτα, Ακούστε και η εξή πρόταση. Να κάνουμε νωρίτερα την επανεξέταση από ό,τι προτείνουμε εμείς. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητούμε να είσαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που ζητάτε. κατά πόσον δηλαδή αυτή η νωρίτερη επανεξέταση θα έχει κάποιο νόημα, κάποια ουσία πρακτικά και κατά πόσον θα μπορέσει να μας επιτρέψει να ορίσουμε νέα μέτρα πολιτικής πέρα από τον ορίζοντα που έχουμε ορίσει πριν το 2030. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, να μην ζητάμε, αν θέλετε, πρόορη υποβολή έκθεσης, γιατί οι προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε ε, σε αυτή την ε, πρόορη, αν θέλετε, έκθεση, δεν θα μας επιτρέψουν να λάβουμε υπόψη ουσιαστικά νέες εναλλακτικέ. Τώρα να επανέλθω σε κάποια επιμέρους ερωτήματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήμουν τόσο ακριβής έως τώρα στα μου, γιατί παραπέμπω στη μελέτη, αλλά σε ό,τι αφορά αυτή τη μελέτη δικτύπου, έγινε με βάση τον υπολογισμό ε, που κάνουμε για τον αντίκτυπο του, ε, προς, τον ΑΕΠ, προς το ΑΕΠ συγγνώμη. και θα είναι 0,009% της, η συνολική δαπάνη στο ΑΕΠ. Χρησιμοποίησαμε δύο μοντέλα υπολογισμού ε, του αντικτύπου στην εργασία και το εν, η μία μέθοδος οδηγεί σε μία αύξηση θέσεων εργασίας κατά 7.000. Ενώ το άλλο μοντέλο υπολογισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ε, 16.000 ε, θέσεων εργασία. Κοντά, κοντά λοιπόν στο 0. Θεωρούμε περιθωριακό αυτό το αποτέλεσμα Και υπάρχουν τομείς στους οποίους σίγουρα προβλέπουμε θετικά αποτελέσματα, να επηρεαστούν γενικότερα θετικά. Και ε, με, με αυτό που προτείνουμε θα υπάρξει αύξηση των μερίδιων αγοράς και διεθνώς για κάποιες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει να επανέλθει κανείς. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειάζεται να επαναλάβω το χρονοδιάγραμμα, κατάθεση τροπολογιών μέχρι τι 26 Απριλίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 30 Μαΐου και ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 19 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν 26 Απριλίου η κατάθεση των τροπολογιών. Στο επόμενο θέμα τώρα, έκθεση του κυρίου Χίγκιν, έκθεση πρωτοβουλία για την η υπηρεσία τηλεδιοδίων και ένα σύστημα αυτοκόλλητων σημάτων για τα ελαφρά οχήματα. Έχει το λόγο. Τζιμ, έχουμε και 59 τροπολογίε. Πρόεδρε, το έχω πει και σε προηγούμενε συνεδρίε για να έχουμε ένα πιο ευθυγραμμισμένο σύστημα και κυρίω επειδή έχουν προκύψει τα προβλήματα στην υπόθεση αυτή. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίω στην μη υλοποίηση, στην μη εφαρμογή των ήδη θεσμοθετημένων ε, νομοθετημάτων. Ευχαριστώ λοιπόν τους κοιόδης ηγητές για την πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε μια πολύ παραγωγική συνεδρία στην προηγούμενη Πέμπτη το πρωί μπορέσαμε να συνενώσουμε σε έξι συμβαστικές τροπολογίες, τις περισσότερες από τις ε, τροπολογίες που είχαν κατευθεί. Ε, η κατάσταση είναι ουσιαστικά ότι οι συμβαστικές τροπολογίες, και το αναγνωρίζω αυτό, ε, έχουν βελτιώσει σημαντικά το αρχικό μου κείμενο. Ως εκ τούτου αυτό που κάνουμε είναι ότι αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ήταν πολύ θετική η συμβολή των σκιωδών εισηγητών και ελπίζω αύριο να στεφθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημα. Ευχαριστώ να συζητήσουμε οποιοδήποτε από τα σχόλια. Κάποια μέλη από ό,τι φαίνεται έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα μόλις έφτασα και δεν πρόλαβα μια συνεδρίαση που είχε ε, προγραμματιστεί και ολοκληρώθηκε πριν από μισή ώρα περίπου. Ε, πάντως αν υπάρχει κάποιος συνάλφος που έχει σχόλιο. Ευχαριστώ. Ναι, και ο κύριο Αλκαντράιερ, ο οποίο τώρα πλέον μεταλλάσσεται σε γυναίκα. Κυρία Γιαλασάντερ, αγαπητέ Αλκαντράουε. Ναι, είναι στο εξωτερικό η κυρία Γιαλασάντερ, Σάντος, ε, πρέπει να το πω. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για τη δουλειά του. Και εμείς βεβαίως θα πρέπει να ε, στηρίξουμε τη γενική προσέγγιση και την πρόοδο στο σύστημα αυτό, το διαλειτουργικό στην Ευρώπη. Πολλή δουλειά ακόμη μένει να γίνει βεβαίως. Τούτου λεχθέντος οι προτάσεις, συμβαστικές προτάσεις του εισηγητή αφήνουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες και ερωτηματικά. Ακόμα μέχρι σήμερα το μεσημέρι έπαιρνα προτάσεις. Τώρα για τις συμβαστικές 1 και 2 αναφέρεται η αναγκαιότητα νέου κανονισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μία λύση, αλλά ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι και άλλες λύσεις για να προχωρήσουμε. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για νομοθετική πρωτοβουλία ή κάποια άλλη πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα την περιφερειοποίηση του συστήματος, εδώ πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να το δούμε σαν ενδιάμεσο βήμα. Διότι πράγματι διασυνοριακά μπορούν να δουλέψουν μεταξύ τους διάφορες χώρες. Θα ήταν ένα διάμεσο στάδιο. Όμως, στο τέλος, θα πρέπει το σύστημα να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Βόρεια μέχρι την Νότια Ευρώπη, να μπορεί κανείς να κυκλοφορεί με ένα σύστημα, με ένα μηχανισμό που να λειτουργεί παντού. Αυτό θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει διάφορα. Συγχρηματοδότηση μέσω του 10-10. να υπάρξει παρετέρω έρευνα. Όσον αφορά τώρα την πρόταση του συγητή για να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα διοδίων που να βασίζεται σε δορυφόρο είναι μια λύση και αυτή, αλλά θα πρέπει να παραμείνει δέτερο το σύστημα. Πάντως εμείς κάνουμε έκκληση να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα που λειτουργεί από απόσταση. Και να γίνει έτσι πιο δίκαιο. Τέλος, για τη συμβαστική 5, εδώ έχουμε την εντύπωση ότι η βασική ιδέα δεν ε, αντικατοπτρίζεται απόλυτα. Και πιστεύουμε επίσης ότι τα κρατημέλη τελικά πρέπει να αποφασίσουν ποιο σύστημα θα εφαρμόζουν. Και τι θα κάνουμε τα έσοδα επίσης. Εμείς θέλουμε τα κράτη-μέλη τα χρήματα τα οποία θα συλλέξουν από το σύστημα αυτό διοδίων να τα επενδύουν σε πιο βιώσιμη κυκλοφορία. Είτε με δρόμους είτε με οτιδήποτε άλλο. Αυτά. Φυσικά και στηρίζουμε τις κύριες γραμμές. Έχουμε βέβαια κάποια ερωτηματικά στους συμβασμού που προτείνονται και θα φροντίσουμε να τους συζητήσουμε παρατέρω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάσινερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εκπροσωπώ εδώ τον Βολφ Κλίντς και ο Δησηγητή ο οποίος θα ήθελε να είναι παρόν αυτοπροσώπος αλλά μια και προχωρήσαμε πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζε στο πρόγραμμα δεν προλαβαίνει να έρθει από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστώ λοιπόν εκ μέρου του τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Χίκινς. Έχουμε συζητήσει το θέμα βεβαίως. Ε, έχει νόημα, είναι σημαντικό, είναι σωστό για χάρη του Ευρωπαίου χρήστη να γίνει εναρμόνιση αυτού του συστήματος ε, τηλεδιοδίων και συστήματος τελών. Κάποια κρατημέλη έχουν εισαγάγει κάποια συστήματα. Για τον, κύριο, για τον κύριο Κλίντς είναι σημαντικό να παραμείνει η δυνατότητα αυτή για το μέλλον, ε, η δυνατότητα της επιλογής δηλαδή για το κράτος μέλος και, για, και έτσι ώστε να γνωρίζει και ο χρήστης ε, να υπάρχει διαφάνεια να ενημερώνεται για το τι προχωρεί στον χώρο των μεταφορών, στις οδικές μεταφορές ε, προσωπικού αλλά και ε, φορτίου στην Ευρώπη. Πρέπει βεβαίως να αξιοποιηθούν μέσα που υπάρχουν όπως το GPS αυτό άλλωστε ισχύει και για τι ε, τηλεαγορέ κτλ. Ο κ. Κλίντ έχει κάνει τη σχετική πρόταση και χαίρεται που έχει αναδεκτεί. Για την περιφερειοποίηση, η κυρία Γιάλα Σέντερ είπε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό βήμα. Είναι σωστή εναλλακτική βεβαίω. Υπάρχουν ε, άλλα συστήματα ε, και έχουμε σε κράτη άλλα τη δυνατότητα μια περιφέρεια να προχωρήσει προς την εισαγωγή του συστήματος και άλλη μη εφόσον δεν το προτιμά. Πάντως, καθοριστικό είναι να γίνει, όπως είπε και ο κύριο Χίγγινς, ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία με αυτό. Κύριε Λίχτινμπέργκερ, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από την αρχή την εισήγηση του κύριου Χίγγινς. Έχουμε στην Επιτροπή των Γυναικών Νομική Επιτροπή και της Νομικής Επιτροπής κοινή ακρόαση για, τα, ε, για την παρουσία των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια. Μη φοβάστε, μη φοβάστε, μη φοβάστε. Είναι ποιοτικέ ε, οι επιλογές. Δεν ναι, ναι, έχετε λόγο να ανησυχείτε. Για το θέμα μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Έκανε πράγματι μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνει και η συζήτηση στους σωστούς όρους στο Στρασβούργο για το θέμα αυτό. Ένα σημείο παραμένει και μενα κάπως κρεμές, γιατί είχα την εντύπωση ότι είχαμε συμφωνήσει πως δεν θα γίνει αναφορά σε κανονισμό. Ωστόσο, βλέπω σε τρεις συμβαστικές τροπολογίες τέτοια παραπομπή. Ίσως θα σκόπιμο να το ξαναελέγξουμε. Εγώ είχα την εντύπωση ότι δεν είχε συμφωνήσει η πλειονότητα των σκιωδών εισηγητών στο θέμα αυτό. Και υπήρχε και το ζήτημα της ε, νομικής ισχύω μιας πρωτοβουλίας τέτοιας, μιας προτάσεως τέτοιας. Γιατί μέχρι στιγμής τίποτε δεν έχει εμποδίσει τα κράτη-μέλη στο να μην εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Άρα θα είχαμε περισσότερες ευκαιρίες για ορθή ε, εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας εάν, ε, αν εισάγαμε κανονισμό. Όπως είπα, η πλειοψηφία δεν έχει υποστηρίξει τη λύση του κανονισμού. Και θα παρακαλέσω το συνάδελφο να το ξανακοιτάξει γιατί έχει σημασία για μένα. Το αν θα παραμείνει η αναφορά ή όχι. Επίσης, Υπάρχουν κάποια ουσιώδου σημασία θέματα, τα οποία βλέπω μέσα στις συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστώ τον εισηγητή. Πάνω απ' όλα, κεντρική σημασία, γιατί η εμπορία που έχουμε συλλέξει αυτό υποστηρίζει, ε, ουδετερότητα ως προς την τεχνολογία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μην χρειαστεί να υποδείξουμε ή να μην καταλήξουμε στην υπόδειξη συγκεκριμένη τεχνολογίας, γιατί αυτό και την καινοτομία πλήττει και εν τέλει είναι μια λύση στην οποία πρέπει ποτέ να καταφεύγει το νομοθετικό όργανο, στην νομοθετική του δράση. Η επιβολή και εφαρμογή της νομοθεσίας έχει εν τέλει τη μεγαλύτερη σημασία για μένα. Η Επιτροπή έμεινε άπραγη μέχρι τώρα ενώ υπήρχαν δυνατότητες στα κρατη με τις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες και εν τέλει δεν έχει μεγάλο νόημα να συζητούμε εις μήκος και εις βάθος όλη αυτή την ιστορία εφόσον εν τέλει δεν προχωρεί η υλοποίηση σωστά. Θα έλεγα ότι αρκετά έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό. Πρέπει πια να απευθύνουμε σαφή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στα δέοντα συμπεράσματα σε σχέση με ορισμένα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα και για τα όσα είπε η κυρία Μάισνερ, ένα αίτημα της κυρίας Αιάλα Σέντερ σχετικό με την περιφερειοποίηση περιφερειακές πρωτοβουλίες. Για μένα δεν είναι πολύ σαφές το σε ποιους τομείς μπορούν πραγματικά να εμφανιστούν αυτές οι περιφερειακές πρωτοβουλίες. Θα, μιλά, θα πρόκειται για ένα σύστημα της αγοράς ε, των ε, τηλεδιοδίων. Ε. Από την άλλη, προκειμένου να μην διονυστεί αυτό το πρόβλημα και να μην χρονίσει, ας ε, βρούμε κάποια λύση η οποία προσφέρει προς αφήνεια. Το έχουμε δει αυτό το πρόβλημα πολλές φορές να παραλαμβάνεται. Και άρα νομίζω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση, να προχωρήσουμε με τους ρυθμούς που μπορεί ο καθένας. Ο κύριος Ζήλα έχει το λόγο. Ο κύριος Ζήλα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια σημεία βέβαια που έχω κάποια διαφωνία, αλλά γενικά εντάξει. Πρώτα απ' όλα όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πιστεύουμε πως η νέα προσέγγιση πρέπει να είναι κανονισμός. Μάλλον οδηγία. Έχουμε δηλαδή την αίσθηση ότι δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν πρέπει να έχουμε δεσμευτικό κείμενο. Ούτε συμφωνώ με την θέση του κειμένου που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν την προτεραιότητα στα συστήματα αυτά που αναφέρονται Σε μερικές περιπτώσεις έχουμε μεγάλα φορτηγά τα οποία κυκλοφορούν μέρα και νύχτα και προκαλούν ζημιές στις χώρες από τις οποίες διέρχονται. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αξιολογούν ποια είναι τα συστήματα εκείνα τα προτιμούν αν είναι της απόστασης του χρόνου. Όσον αφορά την περιφερειοποίηση τώρα, έτσι όπως βλέπουμε εμείς το πράγμα, μπορεί να είναι πιο Η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών διοδίων ίσως θα μπορούσε να πετύχει περισσότερο έτσι. Αντί να έχουμε μία δεσμευτική πρόταση και ένα νέο σύστημα το οποίο στην πράξη να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Ίσως λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε καλύτερα αυτή τη λύση της περιφερειοποίησης. Ευχαριστούμε κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Η γνώμη μου και της ομάδας μου είναι ότι Η πρόταση αυτή κάνει το αντίθετο από την ε, ελευθέρωση. Υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες. Η κάθε μία παίρνει διαφορετικό δρόμο. Όπως είπε και ο κύριος Ζήλερ, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία. Κατά τα άλλα συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Higgins, εξαιρετική δουλειά του. Μία σκέψη, μία ιδέα μόνο. Σε μία θεολογική σκέψη αναφερόμαστε στην αρχή του ε, ο Ριπέρον πληρώνει και νομίζω ότι θα πρέπει ή ο χρήστης πληρώνει. Ε, θα πρέπει να βρούμε κάποια διασύνδεση κάποια αιτιολογική συνάφεια νομίζω. Ίσως ε, στην, στην συμβαστική τροπολογία υπαριθμών πέντε να μπορούσε να εγγραφεί μια τέτοια διατύπωση, για να παραμείνουμε συνεπείς από την αιτιολογική σκέψη στο διατακτικό της συμβαστικής πέντε Κύριε Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη, καταρχάς, που άφησα την κίνδυνο να μιλήσει εκ μέρους μου. Νόμιζα ότι θα αρχίσετε μετά τις 5. Με προλάβατε. Για το άος είπε ο κύριος Κόχ. Βεβαίως και θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε τα έσοδα από, την, ε, από τα τηλεδιώδια να τα αξιοποιούσαμε και για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Συντήρηση κτλ. Πολύ ωραία θα ήταν, αλλά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν μπορούμε εμείς να αγγίξουμε τα χρήματα αυτά. Αλλά σαν στόχο ή σαν επιθυμία ή σαν πρόθεση μπορούμε να το καταγράψουμε. Στη Γερμανία το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για την συντήρηση ούτε καν ε, για βελτίωση του οδικού δικτύου δεν Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Έχουμε μεγάλη δυσκολία ως προς την ε, εφαρμογή στην πράξη των διατάξεων, των νομοθετημάτων που έχουν ήδη εγκριθεί στον τομέα αυτό. Και ως εκ τούτου θα πρέπει και για το μέλλον να επαγρυπνούμε και εδώ η Επιτροπή καλείται να ε, εξασφαλίσει πρόοδο στην υπόθεση αυτή, στην εφαρμογή. Τρίτον, εδώ και χρόνια, μέχρι το 2010, κάναμε είχαμε το στόχο της εξασφάλισης της ε, ε, πρώτης θέσης, της πρωτοκαθεδρίας ε, στην στήριξη της οικονομίας μας στη γνώση. στο της Λισαβόνας, δεν τα καταφέραμε. Το θέμα αυτό λοιπόν, το οποίο συζητούμε, είναι νομίζω ένας από τους τομείς στους οποίους υπάρχει μεγάλο δυναμικό καινοτομία με πολύ πρωτοπόρα δύο. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για να προχωρήσουμε περισσότερο ή να εδραιώσουμε ήδη δοκιμασμένα συστήματα. Διαλειτουργικότητα, ναι, απαραίτητη, δεν υπάρχει φωλία, αλλά ίσως θα ήταν και σκόπιμο να κάνουμε ένα κουαντικό άλμα στην, ή τουλάχιστον να επιδιώξουμε ένα κουαντικό άλμα στην τεχνολογία. Δεν φαίνεται να έχουμε δώσει αρκετή έμφαση στην υπόθεση αυτή. Το πρόβλημα είναι βεβαίως ότι τα κράτη-μέλη που φυλάσσονται του δικαιώματος να αποφασίσουν μόνα τους εάν θα εισαγάγουν σύστημα θεοδίων, τι του σύστημα, εάν θα έχει να κάνει με την χρήση συγκεκριμένων τμήματων του δικού δικτύου, αν θα εξαρτάται από την διανηθήσα απόσταση, και ούτω καθεξής. Καλό θα ήταν να προχωρήσουμε προς ε, πιο ενιαίες προδιαγραφές και πρότυπα και να μην έχουμε πια αυτό το, ε, αυτή την κουρελού με, τα, διαφορετικέ τις διαφορετικές λύσεις που ισχύει στην Ευρώπη. Με πολύ διαφορετικά συστήματα δύο-δύο που εμποδίζουν πολλές φορές και δημιουργούν δυσκολίες και προβλήματα στον χρήστη. Άρα, διαλειτουργικότητα, δυνατότητα προ πληρωμής ή ενδεχομένως προκράτησης, που είναι καλές λύσεις. Και τελευταίο. Θα πρέπει καταρχήν να διασφαλιστεί περισσότερη διαφάνεια για το χρήστη για το τι απαρτίζει, τι εκπροσωπεί το τέλος που πληρώνει, το τέλος των διοδίων, σε τι χρησιμεύει. Αυτά. Πολύ καλή πρόταση του κύριου Higgins, χωρίς προβλήματα, χωρίς διαφωνίες. Μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και στην ψηφοφορία. Στην παραγωγή των συμβαστικών τροπολογιών, για να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περαιτέρω, ώστε να μειώσουμε και των αριθμών ε, των υπόλοιπων τροπολογιών, εκείνων που δεν καλύφθηκαν στις βασικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριος Κάτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Χίγκινς, για τη δουλειά που κάνατε για αυτό το θέμα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για αυτό το φάκελο, Είχα επισημάνει κάποια ε, σημαντικά θέματα, ως θέματα αρχής, ότι πρέπει να πλουστέψουμε τη ζωή μας σε αυτό το τομέα, οπότε σημαντικό είναι όλοι, καθώς ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, να έχουμε ένα νέο σύστημα και όχι κάθε φορά που περνάμε τα σύνορα να πρέπει να καθόμαστε και να στεκόμαστε για να προσπαθούμε να καταλάβουμε το σύστημα. Αν χρειάζεται μια εναρμόνιση σε αυτό το τομέα, κάτι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, σήμερα είναι χαόδες η κατάσταση και θα οξυνθεί το πρόβλημα αυτό γιατί βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται όλο και προστρέφει το κινητόδρομο για τις οδικές μεταφορές και Άρα θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα οξυνθεί περισσότερο στο μέλλον. Αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα και μείνουμε άπρακτοι, τότε στο μέλλον θα έχουμε αντιμετωπίσει μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Έπειτα, να διασφαλίσουμε την ιδιωτική σφαίρα και να γνωρίζουμε καλύτερα το κόστο. Αυτέ ήταν οι γενικέ αρχέ, τι οποίε είχα θέσει εγώ ω προπόθεση για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εν μέρη, ε, πιστεύω ότι έχετε δώσει απάντηση σε αυτές τις αρχές που έθεσα. Το κείμενό σα όμω, θα πρέπει πιστεύω να το ξαναδούμε σε κάποιε λεπτομέρειε. Κύριε Χίγκιν, ε, θέλω να πω ότι λυπάμαι γιατί δεν έχω δει τι τροπολογίε, τι συμβαστικέ. Μόλι τώρα τι είδα και ρωτώ. Η περιφερειοποίηση, κατά μένα δεν είναι απλούστευση, είναι ε, περισσότερο περιπλοκή του συστήματος. Εγώ δεν πιστεύω στην περιφερειοποίηση, εν προκειμένου. Έπειτα, θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Η τροπολογία μου η περίπτωση 22 που μιλά για ευρωπαϊκούς κανόνες χωρίς να αναφέρομαστε συγκεκριμένα ε, στα στοιχεία που έχει συμπεριλάβει στις συμβασικές τροπολογίες, δεν, τα γνωρίζω αυτά. Θέλω να μου το διευκρινίσετε αυτό. Ελπίζω, ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο που να προβλέπει εναρμόνιση για όλους. Τα πράγματα θα είναι όλο και πιο περίπλοκα στο μέλλον. Εγώ δεν ε, πιστεύω ούτε στις βινιέτες ούτε ε, στα σήματα. Εγώ πιστεύω στο σύστημα τη NSS ε, και, και τη χρήση των δορυφόρων, της τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα διαχείρισης πληρωμών που να μην βασίζεται στον χρόνο χρήσης, αλλά στις αποστάσεις. Αυτός που χρησιμοποιεί ε, και δημιουργεί ε, ρήπους θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο. Ο κύριος Καραμίτσος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Χίκινς για την επικοδομητική έκθεση και ευχαριστώ και τα μέλη για τις πολλές τροπολογίες και για όσους ακούστηκαν στη σημερινή συζήτηση. Θα είμαι σύντομος. Κάποιες τροπολογίες ζητούν να εξετάσουμε την ε, προέκταση του, των κανόνων και για άλλες κατηγορίες οχημάτων, εμείς βλέπουμε θετικά αυτή την πρόταση και μπορώ να πω ήδη στην αρχή ότι μπορεί και μέσα αυτή τη χρονιά να κάνουμε μια πρωτοβουλία που να βασίζεται στις αποστάσεις. Επίση, θέλουμε να λάβουμε υπόψη στο μέγιστο βαθμό την ευελιξία για τα κρατημέλη να θέτουν τα τέλη που θα χρεώνουν, ε, εξαιρώντας ε, ενδεχομένως τα τέλη για τη συμφόρηση. Ε, άκουσα και κάποιες παρεμβάσεις που είναι υπέρ της περιφερειοποίησης και της τροπολογίας, ενώ κάποιοι άλλοι διαφωνούν, επιμένουν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη οδό για να έχουμε μια πλήρη ε, ευρωπαϊκή κάλυψη. Για μας αυτός είναι ο στόχος, η πλήρη ευρωπαϊκή κάλυψη και παρακολουθούμε στενά αυτά τα περιφερειακά προγράμματα και να κατά πόσο μπορούν να αποτύσσουν ευρωπαϊκή κλίμακα. Αυτό που μπορούμε να πω νοητικά είναι ότι σε αυτή τη στιγμή ε, στην προκήρυξη που ε, έχουμε βάσει των ευρωπαϊκών δικτύων υπάρχει ένα τέτοιο περιφερειακό πρόγραμμα που καλύπτει σχεδόν το 70% της ευρωπαϊκής επικράτειας. Ελπίζουμε αυτό όμως να μπορέσει να ε, επεκταθεί στο 100%. Αν βεβαίω ε, αξιολογηθεί θετικά. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τροπολογίε, τι οποίε βλέπουμε κάπω προβληματικέ. Δεν ξέρω αν η πρώτη παραμένει στο τελικό συμβαστικό κείμενο, γιατί δεν έχουμε δει τι συμβαστικέ τροπολογίε. Είναι η τροπολογία 14 για το δικαίωμα στου κατόχου των οδών που δεν είναι κάτοχοι, οι ιδιοκτήτε πραγματικά, αλλά να καταβάλουν ένα κατάλληλο ποσό για την χρήση των υποδομών και για τι Υπηρεσίε που συνδέονται με αυτέ. Κάποιοι ανάδοχοι που διαχειρίζονται ε, οδικούς άξονες έχουν ε, αυτό, κάνει αυτό το συνδυασμό και κάποιοι θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων που απορρέουν από οποιαδήποτε υπηρεσία και συναφή την υπηρεσία. Με το λογικό, το σκεπτικό μάλλον ότι αυτέ οι υπηρεσίε έχουν εμπορική αξία μόνο γιατί τα οχήματα τα σε αυτού του δρόμου. Άρα δηλαδή όταν ε, ε, εκεί κοντά υπάρχει ένα ωραίο κάστρο ή ένα πολύ καλό εστιατόριο, θα πρέπει αυτό να δικαιολογεί να λάβει αυτό το μερίδιο. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Μια άλλη προβληματική τροπολογία είναι η υπαριθμό 7, η οποία υπερεκτιμά τις ε, εναπομείνωσες σχολείες. Λίγε είναι οι τεχνικέ προδιαγραφέ που θα πρέπει να βρωθούν σε ό,τι αφορά το GNSS πιο συγκεκριμένα, αλλά είναι ε, ε, ίσονος σημασίας και οι υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές είναι ε, έτοιμες και έχει συμφωνήσει και έτσι για αυτές. Η... Άρα πιο πολύ μιλάμε για τις εφαρμοστικές ε, λεπτομερίες που θα πρέπει να ε, συγκλίνουν για να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα για όλους. Πιστεύω ότι η έκθεση σε αυτό το σημείο διακαθορίζει το θέμα πολύ καλά και αυτή την έννοια πολύ απλά χρειαζόμαστε κάποια συστήματα υπολογιστών να το κάνω αυτό το σύστημα. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι αν ε, με την εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα περιφερειακά, εμείς είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε με μια πρόταση. Όμως είμαστε αισιόδοξοι. Με βάση την τελευταία πρόταση που κάναμε, ε, βλέπουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και ελπίζουμε να έχουμε κάτι αυτό σύντομα. Και να πω ότι Ήδη έχουμε και 22 δικασίες σε παρεμβάσει για τα κράτη-μέλη, δεν θέλω να το πω έτσι με κάπως μαύρο χιούμορ, αλλά 22 ε, ε, προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν έχουν εφαρμόσει τα κράτη-μέλη ορθά την νομοθεσία αυτά για τα που λέτε και εσείς για την παρακολούθηση πρέπει ε, να υπάρχει στενή παρακολούθηση της εφαρμογής. Ευχαριστώ ε, τον κύριο Χίκιν, σε αυτά από μένα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και για όλη την συζήτηση. Κύριο Χίκιν, θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Θα αρχίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόσταση. και πρόσεξα και τα σχόλια για την περιφερειοποίηση. Και ο κύριος Ολικαντροή αναφέρθηκε σε αυτή. Εμείς δεν βλέπουμε την περιφερειοποίηση σαν κάτι τελικό, αλλά σαν κάτι μεταβατικό μόνο. Τώρα για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το δικαίωμα των ιδιοκτητών των δρόμων να πληρώνονται, Συμφωνώ με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει και μια δυσκολία που πρέπει να λυθεί. Εμείς θα προτείνουμε να μην περάσει η τροπολογία αυτή. Όσον αφορά τώρα την τροπολογία 7, Κύριε Κλίνης, εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπατε και για τα συμβαστικά. Το πρόβλημα σε σχέση με το αν θα έχουμε οδηγία ή κανονισμό είναι ότι έχουμε μια οδηγία η οποία έχει λειτουργήσει όσο έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Οπότε τώρα δεν λέμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε κανονισμό, αλλά λέμε ότι θα πρέπει να είναι μία από τις εναλλακτικές που θα έχουμε μπροστά μας και που θα τη χρησιμοποιήσουμε σε τελευταία περίπτωση αν τελικά δεν τα καταφέρουμε με άλλα μέτρα. Για τον κύριο Ελκαντραουή. Αναφέρθηκε και η κυρία Λίτεμπέργκερ και άλλοι είπαν ότι η λέξη κανονισμός υπάρχει στις συμβαστικές τροπολογίες τρεις φορές. Ναι, όντως. Αλλά σαν επιλογή, σαν εναλλακτική λύση, όχι σαν υποχρεωτική λύση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχόλιά σας, τι έχω εδώ, για το τεχνολογικά, τεχνολογικά ουδέτερο σύστημα. Εμείς θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει και να έρθει με προτάσεις. Δεν λέμε ποιο σύστημα είναι καλύτερο από το άλλο. Όχι. Δεν λέμε ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Όχι. Στην κυρία Μέστερ τώρα. Και εκείνα αναφέρθηκε στην περιφερειοποίηση. Επαναλαμβάνω, είναι ε, μεταβατικό στάδιο. Ο κανονισμός πρέπει να δείχνει ότι είμαστε σοβαροί, λέγε η Ντεμπέργκερ, φυσικά. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκριθεί θετικά, τότε θα πρέπει να έχουμε κανονισμό. Μέχρι τώρα είχαμε οδηγία και όχι κανονισμό. Και είδαμε που μας οδήγησε η οδηγία. Συμφωνώ και με τον συνάδελφο Κόκο όσον αφορά την χρήση των διοδίων αυτών. Όλοι συμφωνούμε, θέλουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι η επιβολή, το πώς θα επιβληθεί το όποιο σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Higgins. Αύριο θα ψηφίσουμε. Και έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή μερίσια διάταξη και σε πέντε λεπτά θα συνεδριάσουν οι συντονιστές.